morning, colleagues. Let's start. Καλημέρα συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Καταρχήν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται και Στη συνέχεια έχουμε τον ε, νομισματικό μας διάλογο με τον Μάριο Ντράγκη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ήθελα πραγματικά να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα εδώ. Είναι πάντοτε εδώ στον τακτικό μας διάλογο και εκτιμώ ιδιαίτερος ότι αυτή τη φορά επέλεξε να είναι εδώ ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια πολύ σημαντική διάσκεψη της, των G20 σε επίπεδο κεντρικών τραπεζών και υπουργών οικονομίας ε, στην ε, Αυστρία. Η Αυστραλία. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντράγκη λοιπόν που είστε εδώ για να μας ενημερώσετε για τις νομισματικές εξελίξεις. Ήδη είχαμε την συζήτηση με τους εμπειρογνώμενους του Econ Panel. Εστιάσαμε την προσοχή στις συνέπειες των του μονίμων πληθωριστικών τάσεων. Αναμένουμε εδώ και εσείς να εστιάσετε σε αυτά τα θέματα, διότι αυτή η συνεδρίαση ακολουθεί ε, ε, συμβούλιο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΟ που ανακοινώθηκαν σημαντικά μέτρα. Θα σας δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο να θυμίσω πρώτα τη μέθοδο εργασία μας μετά από μια δεκάλεπτη εισήγηση του κυρίου Ντράγκη. Θα έχουμε ένα πεντάλεπτο για κάθε ερώτηση συμπεριλαμβανομένης της απάντησης και της επιθανής επερώτησης. πρόεδρε Ντράκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή ακρόαση λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή αλλαγών για την ΕΚΤ. Στις 4 Νοεμβρίου η ΕΚΤ θα γίνει ο επόπτης του τραπεζικού συστήματος για την ε, Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εποπτείας 120 μεγάλων τραπεζών. Αυτό σηματοδοτεί το μεγαλύτερο βήμα της οικονομικής, οικονομικής ολοκλήρωσης από την ε, ε, έναρξη του ευρώ. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για το βήμα αυτό, αλλά επίσης γνωρίζουμε την πολύ μεγάλη επιπλέον ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Στη διάρκεια των επόμενων μηνών δε, η πλειοψηφία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μετακινηθούν στις νέους χώρους στο Frankfurt Ostend, ενώ ε, το προσωπικό του, του ενιαίου μηχανισμού εξυγίνησης θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης. Αυτό θα, γεωγραφικά θα υπογραμμίσει το διαχωρισμό ανάμεσα στη νέα εποπτική λειτουργία της ΕΚΤ και των άλλων καθηκόντων της. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δημοσιεύσαμε σήμερα την απόφασή μας για την εφαρμογή του διαχωρισμού ανάμεσα στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και τις εποπτικές της λειτουργίες, όπως αυτό απαιτείται από τον κανονισμό, από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Στις 3 ε, Νοεμβρίου, την παραμονή της έναρξης της ε, ενιαίας εποπτείας, θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε με τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου. Μέχρι τότε, τα αποτελέσματα ε, της συνολικής αξιολόγησης θα έχουν καταστεί γνωστά. Με αυτή τη βάση, σήμερα και στις ακροάσεις από εδώ και στο εξή θα εστιάζω την προσοχή μου στα παραδοσιακά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ιδιαίτερα στην νομισματική πολιτική. Η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη χάνει κάπως ε, την ορμή της. Μετά από κάποιες ε, κάποια ήπια ανάπτυξη της τελευταία τρίμηνα, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη σε πραγματικό ΑΕΠ σταμάτησε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Οι πρώιμες πληροφορίες για τις οικονομικές συνθήκες που λάβαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν κάπως πιο ε, δύναμες από ό,τι αναμενόταν. Ενώ η, μετα... η βιομηχανική παραγωγή και οι παραγγελίες στο μεταπητικό τομέα τον Ιούλιο έδωσαν κάποιες λαβές για αισιοδοξία, πρόσφατες, πρόσφατοι δείκτες δεν, δεν περιλαμβάνουν ενδείξεις ότι η κάθετη πτώση που κατεγράφει τον Αύγουστο σταμάτησε. Στο μέλλον ε, αναμένουμε η εγχώρια ζήτηση να στηριχτεί από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ε, ε, στάση μας στην νομισματική πολιτική, η οποία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, ευνοϊκές ε, χρηματοπιστωτικές συνθήκες, διαθωτικές αλλαγές που στηρίζουν την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Ταυτόχρονα, πολύ ψηλή ανεργία και η διαρκής η ισχνή ανάπτυξη της πίστοσης κάμπτουν την ισχύ της, την ορμή μάλλον της ανάκαμψης. Οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την αναμενόμενη ανάκαμψη είναι μάλλον ε, μεγάλη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γεωπολιτικές συνθήκες ε, που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι κίνδυνοι για ανεπαρκείς ιερωτικές ε, μεταρρυθμίσεις βαραίνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Από το 3% γύρω στα τέλη του 2011 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ε, ακολουθεί καθοδική πορεία εδώ και αρκετό χρόνο. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός εκτιμήθηκε ότι είχε φτάσει στο 0,3% αλλά αργότερα να θεωρήθηκε στο 0,4%. Αναμένουμε ο πληθωρισμός να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες πριν αρχίσει σταδιακά να αυξάνεται το 2015 και το 2016. Δεδομένε της μακρά περίοδου χαμηλού πληθωρισμού που ήδη έχουμε ε, περάσει, θα παρακολουθούμε κινδύνους όσον αφορά τις εξελίξεις για τις τιμές. Ε, ιδιαίτερα θα εστιάσουμε στις πιθανό αντίκτυπο ε, ισχυνού δυναμικού ανάπτυξης, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις εξελίξεις όσον αφορά τις ισοτιμίες, αλλά και το ε, κατά πόσο περνάνε και λειτουργούν μάλλον οι αποφάσεις για την νομισματική πολιτική. Πριν να στραφώ στις τελευταίες μας αποφάσεις για την νομισματική πολιτική, θα ήθελα να τονίσω πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει πάρα πολλά στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών για να ε, προστατεύσει τη σταθερότητα των τιμών. Με επιτυχία καταπολεμήσαμε την κρίση εμπιστοσύνη στο ευρώ που αύξησε τα επιτόκια σε αφύσικα επίπεδα. Προσφέραμε στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης ε, χρηματοδότηση άνευ προηγουμένου και συνεχής, διαρκώς μάλλον ε, χαμηλώναμε τα ποσοστά μας. Ωστόσο, πάνω σε ε, μάλλον με βάση ένα χαμηλό πληθωρισμό και πολύ χαμηλή ανάπτυξη, αποφασίσαμε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να υιοθετήσουμε διάφορες πρωτοβουλίες νομισματικής πολιτικής για να συμπληρώσουμε και να συνοδεύσουμε τα μέτρα που ήδη είχαμε ανακοινώσει τον Ιούνιο. Πρώτον, χαμηλώσαμε το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά 10 βαθμούς ε, στο χαμηλότερο ε, όριο. Το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 0,05% και ε, το επιτόκιο καταθέσεων στο 0,20%. Δεύτερον, ανακοινώσαμε περαιτέρω μέτρα για αύξηση της λειτουργίας της ε, μετάδοσης νομισματικής πολιτικής, στήριξη στην πραγματική οικονομία και δίνουμε, προσφέρουμε περισσότερες νομισματικές διευκολύνσεις επειδή τώρα έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο όριο η αποκατάσταση μιας λειτουργικής ε, μεταφοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά το διατραπεζικό δανεισμό, είναι πολύ βασικό στοιχείο για να εξασφαλίσουμε ότι τα κίνητρα που έχουν ε, εισαχθεί θα φτάσουν στους τελικούς δανειστές και άρα θα στηρίξουν τα πραγματικά εισοδήματα, τις ε, δαπάνες και το σχηματισμό των τιμών. Μετά από αυτή την ανακοίνωση Σύμφωνα με το πρόγραμμά μας για αγορά τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση, το ABS, θα, αγοράσουμε απλούς και, θα, αρχίσουμε μάλλον να αγοράζουμε απλούς και διαφανείς, απλά και διαφανή χρεόγραφα ε, από τον ε, μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα. Επίσης ξεκινάμε την αγορά καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, ε, σύμφωνα με το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων. Ε, επίσης έχουμε την ε, ε, τις στοχευμένες μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης, ε, τα TLTROs, ε, που ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες. Την περασμένη Πέμπτη, 255 τράπεζες συμμετείχαν στην πρώτη τέτοια προσπάθεια αναχρηματοδότησης για ένα ποσό της τάξης των 82,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι εντός της εμβέλειας των αξιών που αναμέναμε με βάση την πραγματική συμπεριφορά των τραπεζών ε, με προηγούμενα προγράμματα. Το Δεκέμβριο οι τράπεζες θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να δανειστούν ε, κονδύλια υπό τη μορφή των αρχικών TLTRO ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να δανειστούν ένα σωρευτικό ποσό ανάμεσα στο Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο 2014 που θα ανέρχεται μέχρι το 7% των ε, δανείων τους στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα με εξαίρεση τα δάνεια για, προς νοικοκυριά για αγορά ακινήτων. Μέχρι το, το, Δεκέμβριο, το Σεπτέμβριο μάλλον και το Δεκέμβριο θα πρέπει αυτά να αξιολογηθούν ε, συνδυασμένα. Από την επόμενη χρονιά θα έχουμε επιπλέον ε, ε, τριμηνία κονδύλια κατά τη διάρκεια των οποίων οι τράπεζες θα μπορούν να έχουν επιπλέον χρηματοδότηση με βάση την απόδοσή τους ε, την δανειοδοτική. Ήδη τα TLTRO έχουν σημαντική θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την αίσθηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, εν γέννη αναμένουμε οι στοχευμένες μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης να λειτουργήσουν σε ένα πολύ στεναρό εργαλείο για να ενισχύσουν την ε, μετάδοση της νομιματικής πολιτικής και να διευκολύνουν νέες ε, πιστωτικές ροές στην πραγματική οικόνομη δεδομένης της δανειακής βάσης της χρηματοπιστωτικής δομής της οικονομίας της Ευρωζώνης θα κατευθύνουμε τα TLTRO σε τρεις κατευθύνσεις. Καταρχήν αναμένουμε τις αγορές απλών και διαφανών ε, τίτλων από τιτλοποίηση με άμεσες επιπτώσεις, δηλαδή το βαθμό στον οποίο η το κόστος της χρηματοδότησης, του δανεισμού, θα ανακουφίσει στις τράπεζες, αλλά θα περάσει και στους ίδιους τους ε, δανειολήπτες, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό να συνδεθεί με τα TLTRO, με με συγκεκριμένο και τρόπο. Ε, αυτό διότι οι δυνατότητες αλλαγής ε, και επιρροής στις δυναμικές των αγορών είναι υψηλές στο συγκεκριμένο τομέα και η σχέση ανάμεσα στα spreads και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ABS στο δευτερεύουσα αγορά αλλά και στα επιτόκια δανεισμού είναι άμεσος και πολύ στενή. Δεύτερον, θα υπάρξει ένα, ένα, μια δίωδος εξισορρόπησης των χαρτοφυλακίων, καθώς η επέκταση της ρευστότητας θα ακολουθήσει τις συνδυασμένες διαδικασίες, καθώς και τη διαφοροποίηση των, ε, των ε, σχημάτων επενδύσεων στην ε, κοινότητα των επενδυτών και άρα θα οδηγήσει σε μια διευκόλυνση των χρηματοπιστωτικών όρων γενικότερα. Τρίτον, πιστεύουμε ότι η γενική νομισματική μας πολιτική υπογραμμίζει την κατεύθυνση και την αποφασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε ε, μια ε, επεκτατική αναπτυξιακή στάση ε, με στόχο τη διατήρηση των, της σταθερότητας των τιμών και τον πληθωρισμό, τη σταθεροποίηση μάλλον του πληθωρισμού κάτω από το 2% μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, η αγορά των ABS αρκεί για να μπορέσουμε να έχουμε μεγάλες αγορές. Οι αγορές μας θα περιλαμβάνουν ένα σχετικά μεγάλο φάσμα απλών και διαφανών ABS που θα είναι εγγυημένα από δάνεια στην πραγματική οικονομία. Το σύνολο των ε, ε, επιλέξιμων χρεογράφων ε, ήδη είναι πολύ σημαντικό. Καθώς και τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα της παρουσίας μας στην αγορά. Με το σύντο χρόνο, καθώς οι αγορές μας θα συμβάλλουν σε μια ομαλοποίηση στις εμπορικές συνθήκες, η δευτερεύουσα αγορά και η έκδοση χρεογράφων θα επεκταθεί και σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι αδρανής. Όπως μας δείχνει η εμπειρία από άλλες κεντρικές τράπεζες, το μέγεθος της αγοράς και η όγκοι αγοράς στην ουσία συναποφασίζονται και είναι ενδογενείς. Οι νέες πρωτοβουλίες τώρα αυτές θα μεγενθύνουν το, την έκθεση σε κίνδυνο του ευρωσυστήματος οι απευθείας αγορές αυξήσουν το μέγεθος ε, του ισοζυγίου της ΕΚΤΑ, αλλά επιπλέον έκθεση σε κίνδυνο θα είναι περιορισμένη. Υπό το πρόγραμμα αγορών ABS αγοράζουμε, μεθαμέν, ε, θα αγοράζουμε νότερες ε, και παλιές μετοχές, μάλλον χρεόγραφα, που είναι ήδη επιλέξιμες για επιχειρήσεις του πράξης μάλλον του ευρωσυστήματος. Έχουμε λοιπόν ευρία εμπειρία όσον αφορά το διαχείριση και την κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτό το τομέα ε, ε, τίτλων. Αυτοί οι τίτλοι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και απλότητα καθώς και από χαμηλούς κινδύνους. Ε, ο μεγάλος βαθμός ανάπτυξης των πιστώσεων που πρέπει να οικοδομήσουν οι βασικοί δανειστές για να προσελκύσουν τα προγράμματα αυτά θα λειτουργήσουν ως ένα περαιτέρω φραγμός κατά των απολειών. Όσον αφορά τις εγγυημένες ενδιάμεσες, ε, ε, τους εγγυημένους τίτλους θα υπάρχει ένας κίνδυνος ο οποίος θα είναι συγκρίσιμος με αυτό του συνεγγυητή είτε σε εθνικό είτε σε υπερεθνικό επίπεδο. Τα καλυμμένα τώρα ομόλογα έχουν κοινά στοιχεία με τα ABS και γι' αυτό είναι συμπλήρωμα στο πρόγραμμα αυτό όπου βάση είναι τα ABS. Η σχέση μεταξύ των δύο είναι σχετικά στενή, καθώς οι τιμές των καλυμμένων ομολόγων αυξάνονται, αναμένουμε οι τράπεζες να ανταποκριθούν στα κίνητα των αγορών και ε, γι' αυτό να υπάρξουν περισσότερα δάνεια ώστε να τα εγγυηθούν. Κατά δεύτερο λόγο, οι άμεσες επενδύσεις σε αυτή την αγορά θα συμπληρώσουν τις αγορές ABS και θα ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια, εξισορροπώντας τις διόδους μετάδοσης και ε, αναζωογόνησης θετικών ε, ε, κινήσεων στις άλλες αγορές και στα ε, χρεόγραφα ή τους τίτλους. Συνδυασμό των μέτρων που ανακοινώθηκαν ανάμεσα στον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο θα έχουν μεγάλη, μεγάλη επιρροή όσον αφορά το ισοζύγιο της ΕΚΤ που αναμένεται να κινηθεί προς τις διαστάσεις που είχε στις αρχές του 2012. Με αυτά τα προγράμματα αγορών ξεκινάμε μια μετάβαση από, μια νομισματική, από ένα πλαίσιο μάλλον νομισματικής πολιτικής που βασικά ε, στηριζόταν στις παθητικές ε, παροχές μιας ε, πίστοσης από την Κεντρική Τράπεζα σε πιο δραστήριο και έλεγχο και διαχείριση του ισοζυγίου μας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους ε, από το μεσοπρόθεσμο η κατάσταση του πληθωρισμού και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μη συμβατικά μέσα εντός των εντολής και να αλλάξουμε το μέγεθος και τη σύσταση των μη συμβατικών παρεμβάσεών μας αν αυτό καταστεί απαραίτητο ώστε να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω κινδύνους ε, μιας μακράς περίοδου χαμηλού πληθωρισμού. Ωστόσο να προσθέσω πως η επιτυχία των μέτρων μας βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που είναι εκτός της νομισματικής πολιτικής, ε, θαραλές διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, βελτιώσεις της ανταγωνιστικότητας ε, του επιχειρηματικού τομέα είναι πολύ βασικά για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό θα παροτρύνει τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε επιγόντως και θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ζήτηση για πιστώσεις. Οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις θα συμπληρώσουν την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και θα ε, διαδώσουν περισσότερο αυτή την ε, νομισματική πολιτική και τα, τις επιπτώσεις της. Όπως έχω πει επανειλημμένα, καμία νομισματική ή οικονομική πολιτική δεν έχουν νόημα χωρίς τέτοιες ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Η κρίση θα τελειώσει μόνο όταν θα αποκατασταθεί πλήρη εμπιστοσύνη στην πραγματική οικονομία και όλο ιδιαίτερο στη δυνατότητα και η προθυμία των εταιριών να αναλάβουν κινδύνου, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση. Αυτό εξαρτάται από μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων συμπεριλαμβανομένη τη νομισματική μα πολιτική, αλλά επίση και ίσω ακόμη πιο σημαντικό είναι η εφαρμογή των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων που στηρίζουν την αξιοπιστία του οικονομικού πλαισίου και την ενίσχυση Τη της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Αρχικά είχατε επίση επιλέξει τις ε, διαφοροποίησης πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ως ένα από τα θέματα της σημερινής ακρόασης. Ελπίζω να κατανοήσετε ότι δεδομένων των σημαντικών αποφάσεων που λάβαμε τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο εστίασα τις παρατηρήσεις μου στα μέτρα νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, είμαι φυσικά έτοιμος και ενδιαφέρομαι πολύ να συνεχίσω να, να συζητήσω μαζί σας το θέμα της επιμονής αυτού του πληθωρισμού που συνδέεται με την ατζέντα των, μεταρρυθμ, των μεταρρυθμίσεων, των, με, διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παύλο Ζάλπα, τον πρώτη μας ομιλητή από το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε Ντράγκη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σα αυτή στην Επιτροπή και ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα κάπως καθυστερημένα και δεν άκουσα την ομιλία σας από την αρχή. Θα ήθελα να μιλήσω για την πρώτη δημοπρασία των TLTRO, των στοχευμένων μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρηματοδότηση. Είπατε ότι ε, δεν διαψεύστηκαν οι προσδοκίες. Ε, βέβαια είπατε ότι η αγορά είναι κατακαιρματισμένη, δεν υπάρχει καλή διαβίβαση και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτή τη φορά οι τράπεζες είχαν την ευκαιρία για φθηνό δανεισμό. Ο κίνδυνος όμως αποφεύγει, ε, α, εμποδίζει μάλλον, τους εμποδίζει να δανείσουν περαιτέρω αυτά τα χρήματα που οι ίδιες οι τράπεζες δανείστηκαν με χαμηλά επιτόκια το φθηνό χρήμα που έλαβαν δεν μπορούν λόγω του κινδύνου να το δανείσουν περαιτέρω. Αυτή ήταν λοιπόν αυτός ήταν η πρώτη δημοπρασία ρευστότητα, ο πρώτος πληστηριασμός και μάλιστα έγινε πριν την διεξαγωγή των δοκιμών αντοχής για τις τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλήσατε για μια ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική που θα ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ επίσης ότι χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η νομισματική πολιτική δεν θα μας εξυπηρετήσει καθόλου ή θα μας εξυπηρετήσει ελάχιστα. Τώρα υιοθετείτε μια πιο δραστήρια νομισματική πολιτική. Αυτό το κάνετε γιατί πιστεύετε ότι οι χώρες είναι πιο έτοιμες, πιο και πρόθυμες να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Η Ισπανία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα από τις χώρες ε, που εφάρμοσε τις περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτύσσεται με τους ε, οργότερους ρυθμούς και δημιουργεί και θέσεις απασχόλησης. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια τάση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πολύ πιο ισχυρή από ό,τι στο παρελθόν. Και γι' αυτό εσείς ε, τη συνδυάζετε αυτή τη διαφορά με μια πιο δραστήρια νομισματική πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για την πρώτη ερώτηση. Πρόσφατα είδαμε κάποια σημάδια πολύ περιορισμένης βελτίωσης. Είδαμε δηλαδή ότι ήταν ε, χαμηλότερη η ταχύτητα της ύφεσης. Ωστόσο η τελευταία έρευνα δείχνει ότι οι πιστοτικές προδιαγραφές έχουν μετριαστεί σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα δανεισμού τραπεζών και δείχνει επίσης ότι παρότι είναι πιο αυστηρές, ότι παραμένουν πιο αυστηρές προδιαγραφές από ό,τι πριν το 2003 ιστορικά. Υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Επί παραδείγματι ρωτούμε τις τράπεζες ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι εμποδίζουν την διαδικασία ε, του δανεισμού από πλευράς της προσφοράς και η απάντηση πολύ συχνά ήταν η αντίληψη για τον κίνδυνο, δηλαδή η προσπάθεια αποφυγής του κινδύνου. Αυτός ο παράγοντας έχει περιοριστεί στις τελευταίες έρευνες. Αλλά οι πιστοτικές προδιαγραφές παραμένουν οι ίδιες με την ε, αρχική εκείνη περίοδο του 2003. Απλώς δεν βλέπουμε γιατί δεν αναπτύσσονται οι τράπεζες. Μας λένε ότι εάν έχουν τη δυνατότητα θα συνεχίσουν να προσφέρουν ε, συνθήκες χρηματοδότησης με πολύ πολύ καλά ε, συνθήκες και για περίοδο μακρύτερη αυτή που αρχικά είχαν προβλέψει, δηλαδή όταν ε, πρωτοαναγγείλαμε τον Ιούνιο τα μέτρα αυτά. Άρα όταν μπει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα θα υπάρχει επαρκέστατη χρηματοδότηση. Κάτι άλλο που διαφοροποιεί TLTRO σε σχέση με προηγούμενες δραστηριότητες που είχαμε αναλάβει τον, ε, το 2012 ήταν ακριβώς το γεγονός ότι αυτά στοχεύουν στην χρηματοδότηση του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα. Οι πρώτες δραστηριότητες του 2012 είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ε, χρηματοδότησης το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ σημαντικά και μεγάλη σειρά ατυχημάτων τραπεζικών που χάρη στα TRO μπορέσαμε να αποφύγουμε το 2012. Τώρα όμως συνθήκες είναι διαφορετικές. Έχουμε συνθήκες χρηματοδότησης επαρκέστατες, αλλά δεν βλέπουμε να διοχετεύονται ή δεν διοχετεύονται επαρκώς ή πλήρως εκεί που θέλουμε, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα. Ε, άρα μπορούμε να προσφέρουμε έτσι πολύ καλές συνθήκες για τις τράπεζες που θα προσφέρουν δανεισμό στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να μην επιδιώκουν άλλου τύπου επενδύσεις με τα χρήματα αυτά. Και κάτι ακόμη για την νομισματική πολιτική. Είναι εδώ κάτι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής. Έχουμε για την ε, αποκατάσταση εμπιστοσύνη ε, την νομισματική πολιτική βέβαια, τις μεταρρυθμίσεις τριαρθρωτικές ε, και την οικονομική πολιτική που θα, θα ακολουθήσει. Αλλά εδώ δεν έχουμε να πούμε κάτι σαν προϋπόθεση ότι η νομισματική πολιτική μόνο εφόσον γίνει αυτό και εκείνο μπορεί να αποδώσει. Δεν υπάρχει ζήτημα δηλαδή διαπραγμάτευσης εν προκειμένου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε εντολή η εντολή μας είναι να διατηρήσουμε το ποσοστό του πληθωρισμού κάτω από το 2%. Ευχαριστώ η Ελίζα Φεραίρα, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά αυτή τη φορά για να είμαι πιο γρήγορη. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σας προσωπικά για το ρόλο της ΕΚΤ στη διάρκεια της κρίσης αλλά και μετά την κρίση. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το ρόλο σας, γιατί ξεκινήσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι θα είστε η εποπτική αρχή στην Τραπεζική Ένωση και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Η ΕΚΤ όμως ε, είχε αναμειχθεί στενά και στον ε, στην εποπτεία των πιο σημαντικό, ε, στις πιο σημαντικές τράπεζες της Πορτογαλίας στα πλαίσια της Τρόικας και τέσσερις ε, μήνες μετά το πρόγραμμα μια μεγάλη τράπεζα της Πορτογαλίας, η του Σάντου, κατέρευσε με τεράστιο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και στη γενική χρηματοπιστωτική σταθερότητα της πατρίδας μου. Τι πήγε στραβά λοιπόν, ποιος ήταν ο ρόλος σας στη Δρόικα. Μήπως τώρα έχετε την αίσθηση ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον εποπτικό της ρόλο στο μέλλον για το ρόλο της ενίας εποπτικής αρχής που θα αναλάβει στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να μας διαφωτίσετε με κάποια σχόλια για το τι συνέβη κατά τη γνώμη σας, τι πήγε στραβά. Επίσης ε, ε, νομίζω ότι ήταν πολύ αξιοσημείωτη αυτή η ένεση ρευστότητα στην Ευρωζώνη από την ΕΚΤ. Αυτή η ρευστότητα όμως ε, δεν είναι και πολύ ρευστή. Δεν πηγαίνει δηλαδή στην πραγματική οικονομία. Και ίσως ήταν ανεπαρκή κοινή στόχη για τα TLTRO, τις στοιχευμένες μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης. Ερωτώ λοιπόν, είναι δυνατόν να έχει εργαστεί κανείς τόσο σκληρά και τόσο άοκνα στην νομισματική πολιτική χωρίς να έχει την αναμενόμενη αντίδραση από τις πολιτικές που θα επηρεάσουν θετικά την πραγματική οικονομία και θα την προσετεριστούν, θα την προσελκύσουν ώστε να λάβει μέρος. Μήπως πιστεύετε ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να γίνουμε όλοι πιο κατηγορηματικοί και πιο ρητοί και να ζητήσουμε μια αλλαγή στο οικονομικό πρόγραμμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Και πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Χώρες που έχουν πλεόνασμα όπως η Γερμανία να αλλάξουν την πολιτική τους. Ή μπορούμε να αρκεστούμε μόνο και να στηριχτούμε μόνο στην επένδυση. Γιατί η προσφορά, στον τομέα της προσφοράς έχουμε καταβάλει προσπάθειες, αλλά δεν είχαμε πάρα πολλά αποτελέσματα. Ποια είναι η πρότασή σας λοιπόν. Ευχαριστώ. Για την πρώτη σας ερώτηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ακόμη ο επόπτης αυτών των τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είχε εποπτικές εξουσίες επί των πορτογαλικών τραπεζών ή επί οποιοδήποτε άλλη τράπεζας. Αυτές τι εξουσίες θα τις αναλάβει από τη στιγμή που γίνει ενιαία υποπτική αρχή. Οπότε η συμμετοχή της ΕΚΤ ε, στην κατάρρευση τη Εσπίρη του Σάντο περιορίζεται στη συμμετοχή της στα πλαίσια της Τρόικα. και δεν είχε σχέση με τη συγκεκριμένη τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άσκησε ε, μάλλον έδωσε στην εποπτική αρχή της Πορτογαλίας καλύτερες ε, προδιαγραφές και συνέβαλε στις προσπάθειες της Τρόικα στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση καλύτερων προδιαγραφών, καλύτερων ε, αναλύσεων της, του δανεισμού. Και χάρη σε αυτές τις καλύτερες προδιαγραφές, η, Ευρωπαϊκή, η Πορτογαλική συγγνώμη, η Εποπτική Αρχή ε, κατάλαβε και το θέμα του BS. των καλύτερων δηλαδή προδιαγραφών ε, του δανεισμού. Φυσικά, εμείς προσπαθούμε να τηρήσουμε την εντολή μας, δηλαδή να κρατήσουμε τον πληθωρισμό γύρω ή κάτω από το 2%. Και αυτό είναι δύσκολο ακόμη και στην παρούσα κατάσταση. Βέβαια, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο ε, σκοτεινή όπως φαίνεται. Γιατί πολλές χώρες έχουν ε, σημειώσει πρόοδο και ήδη αρχίζουμε και δρέπουμε τους καρπούς και βλέπουμε κάποια θετικά αποτελέσματα από τις ε, μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσαν οι, τράπεζες, οι χώρες συγγνώμη, την τελευταία διετία. Πάντως, θα πρέπει να έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για την νομισματική πολιτική μας για να είναι η νομισματική πολιτική μας αποτελεσματική. Και πέραν των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που είναι πολύ σημαντικές, ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η δημοσιονομική πολιτική. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στο Jackson Hall. Η δημοσιονομική πολιτική έχει πολλές διαστάσεις. Έχουμε καταρχήν δημοσιονομικούς κανόνες με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και η υπονόμευση των κανόνων αυτών ισοδυναμεί με υπονόμευση της εμπιστοσύνης. Θυμάστε πώς ήταν η δημοσιονομική κατάσταση πριν από 4-5 χρόνια. Πάντως υπάρχουν κάποια περιθώρια. Υπάρχει και εντός του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εντός των καντώνων τους υπάρχει περιθώριο για κάποια ελαστικότητα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Και να πω και εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει και να αξιολογήσει αυτούς τους κανόνες. Πάντως γενικώ οι χώρες που δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών, τι μπορούν να κάνουν. Καταρχήν, μπορούν να δουν το θέμα της ελαστικότητας, αλλά ποιο είναι πιο σημαντικό για αυτές. Είναι να θέσουν νέες προτεραιότητες, να τροποποιήσουν την ιεράξη των προτεραιοτήτων τους στη δημοσιονομική τους πολιτική εφαρμόζοντας μέτρα δημοσιονομικής εξυγίαση που θα είναι φιλικά προς την ανάπτυξη. Θα δώσουν περισσότερη προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις, στη μείωση των φόρων και θα δώσουν λιγότερη έμφαση σε κάποιες αντιπαραγωγικές και αναποτελεσματικές κρατικές δαπάνες. Βέβαια, και χώρες που δεν έχουν πολύ περιθώριο δημοσιονομικό ε, θα καθοριστούν από αυτούς δύο δρόμος που σας είπα. Τώρα, οι χώρες που έχουν περιθώριο ε, δημοσιονομικό θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ειδικέ συστάσεις χώρα που εγκρίθηκαν από όλους τους ηγέτες ε, των Ευρωπαϊκών χωρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των στρατικών μεταρρυθμιστών, ο κύριος Πέρντς Λούκιν. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Τράγκη, Ήδη και εσείς αναφέρατε το πρόβλημα του κινδύνου του αποπληθωρισμού. Είναι ένας από τους κινδύνους που θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ένας κίνδυνος... Με ακούτε? Τώρα ναι. Λοιπόν, αναφερθήκατε και εσείς ο ίδιος στο πρόβλημα του στον κίνδυνο του αποπληθωρισμού είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα πρέπει να λάβουμε υπόψη για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τους. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το εξής ερώτημα. Μια και είναι χαμηλά τα επίπεδα του πληθωρισμού και υπάρχει ήδη ένα ενδεχόμενο αποπληθωρισμού και μια και δεν έχουμε προχωρήσει πολύ τα τελευταία τρία χρόνια στα μέτρα M3 που θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει μετά την διεύρυνση του M1, νομίζω ότι τα ποσά του M1 θα πρέπει να διαφοροποιηθούν από τα ποσά του M3 σε περίοδο αποπληθωρισμού, δηλαδή τη δυνατότητα περιορισμού των ποσών που μπορεί να έχουν ε, αρνητικά, αρνητικές συνέπειες. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε σε σχέση με τα ποσά αυτά και τι μπορείτε να πείτε σε σχέση με πολύ διστακτικές τάσεις ορισμένων επενδυτών στην διάθεση ε, ρευστότητας προς τις τράπεζες ακριβώς επειδή υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα γιατί βλέπουμε ότι επενδύουν σε, άλλους, σε άλλα επενδυτικά αγαθά, μετοχές και το καθεξής οι τράπεζες, αλλά δεν επιλέγουν επενδυτικά στοιχεία της κατηγορίας M3. Γι' αυτό λοιπόν με το EBS, ε, e με τα EBS ή με τα TLTRO μάλλον δεν λύνει το πρόβλημα γιατί πάνω απ' όλα πρόκειται για ένα πρόβλημα εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα. Θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Όντως, τα M3 έχουν ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης χαμηλό, συμφωνώ απολύτως, για αρκετό καιρό τώρα. Αν και τον Ιούνιο βλέπουμε να έχουν μια μικρή αύξηση, 1,6% έγινε 1,8%. Τα M1 τώρα είναι τα μόνα τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της κατηγορίας M3 ουσιαστικά πάλι χωρίς σημαντική ενίσχυση αλλά από το 2,5 του 2,4 του Ιουνίου πήγε στο 2,5 τον Ιούλιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια αυτό είναι η άλλη όψη θα έλεγα των ε, ασθενών ροών πιστώσεων που διαπιστώνονται στο τραπεζικό τομέα. Γιατί είναι από τη μία περιορισμένη η προσφορά ή και η ζήτηση. Θα μπορούσε αυτό να οφείλεται λοιπόν σε μια περιορισμένη προσφορά γιατί έχουν ασθενείς κεφαλαιακές θέσεις οι τράπεζες και ως εκ τούτου περιορίζουν την πίστοση που διαθέτουν γιατί δεν έχουν αρκετό κεφάλαιο. Σε ένα βαθμό Πολλά γίνανε τον τελευταίο χρόνο, τελευταίους 18 μήνες, από τη στιγμή δηλαδή που ανακοινώσαμε ότι πριν αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη ως εποπτική αρχή, θα προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση ποιότητας ε, ενεργητικού και ε, δοκιμής αντοχής, stress test. Και η πρώτη αντίδραση ήταν η άντληση κεφαλαίων. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη γιατί έγιναν νέες πρωτοποριακές επιλογές προς την άντληση κεφαλαίων τους τελευταίους 18 μήνες. Ταυτόχρονα είναι αρκετά πιθανό βράχη πρόθεσμα η αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού και το τεστ αντοχής να οδήγησαν από μόνα τους σε μια μικρή συστολή-περιστολή των ρο, κεφαλαιακών ροών γιατί οι τράπεζες ήθελαν να είναι έτοιμες να έχουν καλά αποτελέσματα ως προς το τεστ αντοχής και ίσως αυτό ακριβώς να οδήγει στα, στα χειρότερα αποτελέσματα. Ποια είναι η εναλλακτική δηλαδή θα έλεγα σε μια τελευταία ανάλυση. Εάν είμαστε πεπισμένοι ότι ε, ε, νοσούν οι τράπεζες, αν έχουν ε, μη αποδοτικά δάνεια στο ισοζυγείο τους, χωρίς εμείς να αναλάβουμε δράση, θα μετα, τις μετατρέψουμε σε τράπεζες ζόμπι, όπως είδαμε να συμβαίνει στην Ιαπωνία, γιατί ούτε θα δανείζουν, ούτε θα δανείζονται. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια πληγή, ένα τραύμα που πρέπει να απολυμανθεί αμέσως, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα οδηγήσουμε σε περισσότερη αιμορραγία. Αλλά με την απολύμανση αρχίζει σιγά σιγά και η ίαση και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε τράπεζες με πιο ισχυρές θέσεις, με πιο στεναρές θέσεις. Από αυτή την έποψη λοιπόν εμείς δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα ως προς την εισαγωγή ενός προ προγράμματος TLTRO ή ABS. Γιατί από τη στιγμή, ιδιαίτερα με το ABS, ε, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα, σταματάει λίγη το AQR και τα τεστ αντοχής. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης μεταξύ των δύο. Ακόμα όμως και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Εμείς ως ε, απόφαση νομισματικής πολιτικής πρέπει να αντιλάβουμε την απόφαση αυτή. Δεν μπορούμε να εσωτερικεύσουμε τις ε, ιδέες ή τις όποιες σκέψεις περί εποπτείας και συνοποιών αυτής αναμειγνύοντας τους δύο τομείς. Αυτό αφορά, όπως είπα, την προσφορά. Ξέρουμε όμως επίσης ότι η επέκταση του δανεισμού περιορίζεται και λόγω της ζήτησης. Και γι' αυτό είπα στο τέλος της αγωγικής μου παρέμβασης ότι μόνο όταν επανέλθει η εμπιστοσύνη για τον τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, μπορούμε να περιμένουμε όταν δηλαδή υπάρχει διάθεση να λάβει κάνει κίνδυνο και να ε, δημιουργήσει νέες θέσεις εργασία. μπορούμε να δούμε μια ανάκτηση, ανάνυψη αυτής της ζήτησης. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο στο οποίο, σαν πρώτο βήμα, θα επανέλθει η εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ εκ μέρου των φιλελευθέρων Ραμών Τρεμόσα Ιμπάλσα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας ε, αγαπητέ πρόεδρε Ντράκη και καλώς ήρθατε και πάλι. Θα κάνω την ερώτησή μου στα αγγλικά. Αγαπητέ Πρόεδρε, πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον Νότο, δεν έχουν πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό. Και μάλιστα αναγγείλατε πρόσφατα το πρόγραμμα αγορά τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση, τον ABS. Μήπω όμω οι τράπεζε δανείζουν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει όχι επειδή φοβούνται την αφαιρεγκαιότητα, αλλά επειδή είναι υψηλά τα τέλη δανεισμού ή τα, τα επιτόκια δανεισμού και πιστεύετε ότι τα υψηλά, οι υψηλές χρεώσεις του δανεισμού είναι, αποτρεπ, είναι έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για το δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από πλευρά τραπεζών. Πιστεύετε αν μειωθούν τέτοια, τέτοια βάρη στο κεφάλαιο ε, για το δανεισμό προ τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αυξηθεί η πιστοτική ροή προ αυτέ. Ευχαριστώ. Σίγουρα διαπιστώνουμε ότι και οι όγκοι αλλά και οι όροι και προϋποθέσεις στη δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι υψηλότεροι από άλλες μορφές δανεισμού. Διαπιστώνουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιτοκίων ε, δανεισμών ε, μεγάλων επιχειρήσεων και των επιτοκίων δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Φυσικά υπάρχουν και διαφορές ε, μεταξύ των χωρών στα επιτόκια αυτά. Και η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών δανειοληπτών υπήρχε ανέκαθεν. Δεν είναι κάτι καινοφανές. Βέβαια, η διαφορά σήμερα έγκυται στην διεύρυνση, στην μεγάλη διαφορά των επιτοκίων που είχε αυξηθεί το 2012, άρχισε να πέφτει το 2013 και τώρα έχει μειωθεί αυτή η διαφορά μεταξύ επιτοκίων προς δανεισμού μεγάλων επιχειρήσεων και επιτοκίων δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι πολλές επιχειρήσεις επέστρεψαν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά είναι χρονοβόρα η διαδικασία ανάκτησης της εμπιστοσύνης προκειμένου να την, να δούμε, να την δούμε απτά και στην πραγματική οικονομία. Πάντως και οι διαφορές στον όγκο δανεισμού είναι μεγάλες. Και για τις διαφορές αυτές υπάρχουν δύο-τρεις λόγοι. Πολύ συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν χαμηλότερο, μικρότερο κεφάλαιο ε, και λαμβάνω συνήθως περισσότερη μόχλευση από τις μεγάλες επιχειρήσεις, από τους μεγάλους ομίλους εταιριών. Και στις συγκρίσεις αυτές θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι και ολόκληροι τομείς έχουν εξαφανιστεί σε αυτή την αναδιάρθρωση που έγινε της οικονομίας μας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τέτοιους τομείς έχουν εξαφανιστεί, μια και έχει εκλείψει ο ίδιος ο τομέας. Για παράδειγμα στον οικοδομικό τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα, που έχει καταβαραθρωθεί σε μία-δύο χώρες. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του κινδύνου. Και σίγουρα μεγάλος, ε, μεγαλύτερο κίνδυνο έχει μία τράπεζα όταν δανείζει σε μικρομεσαία επιχείρηση από όταν δανείζει σε μεγάλο εταιρικό όμιλο. Και από την έρευνα τραπεζικού δανεισμού έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η αντίληψη του κινδύνου έχει μειωθεί αισθητά το τελευταίο 1,5 χρόνο και έτσι πειράζει λιγότερο την παροχή δανεισμού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίζα Ματίας, εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντράγκη για την παρουσία σας. Πριν από ένα μήνα είχατε έρθει και πάλι στην Επιτροπή και κάνατε δηλώσεις που αν τις παίρναμε σοβαρά θα είχαν ανατρέψει την κατάσταση στην Ευρώπη. Γιατί είπατε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τη λιτότητα και να προσανατολιστούμε στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν με εντυπωσίασαν ούτε οι προηγούμενες δηλώσεις ούτε οι σημερινές. Γιατί δεν βλέπω καμία διαφορά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το να λαμβάνει υπόψη αυτές τις δηλώσεις σας. Όλα τα μέτρα που αναγγείλατε ουσιαστικά ενισχύουν την προσφορά και όχι τη ζήτηση. Γιατί στη ζήτηση έχουμε πρόβλημα και παρόλα αυτά δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και τα μέτρα που αναγγείλατε δεν είχαν καμία, και μέχρι, τα μέχρι τώρα μέτρα δεν είχαν καμία θετική επίπτωση ούτε στην πραγματική οικονομία ούτε στις επενδύσεις. Δεν είναι ότι διαφωνούμε με μη συμβατικά μέτρα ή με χαμηλά επιτόκια. Καλά είναι αυτά τα μέτρα. Πάντως η ρευστότητα χωρίς δημόσιες επενδύσεις θα, δεν θα οδηγήσει πουθενά και έτσι τα μέτρα θα μείνουν αποτελεσματικά και στο μέλλον. Γιατί ο φιλελεύθερος φανατισμός είναι το αδύνατο σημείο της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυτός δυστυχώς κυριάρχησε στους διάφορους θεσμούς μας και δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στον δρόμο επένδυσης και ε, απασχόλησης και ανάπτυξης. Έχουμε αιμονή στο χαμηλό πληθωρισμό απλώς. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη αφορά την δημοσιονομική ελαστικότητα. Ερωτώ λοιπόν, αυτή η δημοσιονομική ελαστικότητα που αναφέρατε, που υπενηχθήκατε, μπορεί να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών δημοσιονομικό και χαμηλό, δανεισμό, ε, χαμηλό ε, κόστος δανεισμού στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή η ελαστικότητα αυτή απλώς θα χρηματοδοτήσει τις δημόσιους υπαλλήλους και θα αυξήσει ουσιαστικά την ανεργία. Είστε έτοιμος ε, να συμβάλλετε ώστε να μειωθεί και το κόστος χρηματοδότησης των χωρών. Είστε έτοιμος να συμβάλλετε ενεργά στο να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των χωρών μελών μέσω της ε, χορήγησης ε, τραπεζικής άδειας στο μηχανισμό σταθερότητας ή μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Uh, Τα μέτρα μας, όπως είπατε, λειτουργούν ε, στο να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια στον ιδιωτικό τομέα σε χαμηλό, με χαμηλότερα επιτόκια. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το 80% της ε, πιστοτικής διαμεσολάβηση στον Ευρωζώνη περνά από την ε, τραπεζική δανειοδότηση. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έτσι λειτουργεί η οικονομία μας. Αν λοιπόν θέλαμε να επεκτείνουμε τις πιστώσεις, πρέπει να περάσουμε από τις τράπεζες. Και η πρώτη προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε για να παρακάμψουμε τις τράπεζες, αν και θα παραμείνουν σημαντικέ, ακριβώς είναι είναι η εισαγωγή του προγράμματος ABS, τίτλων από τίτλοποίηση, αγοράς τίτλων δηλαδή. Δεν είμαστε, όπως είπα, που μόνο το 30% της πιστοτικής διαμεσολάβησης γίνεται μέσω των τραπεζών. Επόμενη παρατήρηση είναι πώς θα μπορούσε η ΕΚΤ να βοηθήσει, να στηρίξει τους προϋπολογισμούς των, ε, τους κατοικούς. Αυτό δεν είναι δικό μας έργο, δεν είναι στην εντολή μας αυτό. Και μπορώ να πω και κάτι παραπάνω, ότι είναι τελείως εκτός της εντολής μας. Αλλά εάν ε, δείτε τις εντυπωσιακέ αποταμιεύσεις που μπόρεσαν να κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις λόγω της νομισματικής, των νομισματικών αποφάσεων της ΕΚΤ που τις έλαβε έχοντας μόνο υπόψη την σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να διερωτηθείτε. Πού πήγαν αυτές οι αποταμιεύσεις, πού πήγαν, σας ρωτώ εσάς. Οι νέε λοιπόν προτεραιότητες σε συνιστώσεις του προϋπολογισμού εδώ είναι πολύ σημαντική. Αυτό που συνέβη στους κατοικούς προϋπολογισμούς από το 2012 και μετά ήταν ότι σημαντικά ποσά εξοικονομήθηκαν από τις πληρωμές ε, για την εξυπηρέτηση των χρεών, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν ε, για αυτούς τους στόχους και σε ορισμένε χώρες μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν για καλά προγράμματα που απέδωσαν ε, κέρδη ενώ σε άλλες χώρες χρησιμοποιήθηκαν απλά για να ε, καλύψουν τις τρέχουσες δαπάνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η πράσινη Σφεν Κίγκολτ. Πρόεδρε Δράκη. Οι προτάσεις των τεσσάρων προέδρων και οι δικές σας προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης είναι αποκρισταλωμένες πια και έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετούς εκπροσώπους κυβερνήσεων που συναντιούνται στη Γερμανία με τον κύριο Βάλς ε, σε συνεντεύξεις τύπου που είναι πολύ δύσκολο να ακούσει κανείς. Δεν βλέπουμε κανένα σχέδιο μεγάλο παρά την κρίση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και μας πικραίνει πολύ το να δούμε ότι είναι τόσο, το, το να δούμε ότι είναι τόσο περιορισμένα τα κίνητρα για την αναζωγόνηση της οικονομίας. Βλέπω λοιπόν ότι είσαστε υποχρεωμένος να ε, προσπαθήσετε με εμβαλωματικές λύσεις να βοηθήσετε την Ευρωζώνη. Τα LTRO στο παρελθόν αγόραζαν κρατικά ομόλογα για να μπορέσουν να ε, διευκολύνουν τη ρευστότητα στην αγορά και να αποκαταστήσουν κάπω την εμπιστοσύνη. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω το εξή ενώ σε αυτή τη κατάσταση Προσπαθήσατε ποτέ να προσμετρήσετε πόσο υψηλά ήταν τα κέρδη τα οποία αποκόμισαν οι τράπεζε από αυτό το carry trade. Και δεύτερον, θα μπορούσατε να μας δεθέσετε τα στοιχεία αυτά. Δεύτερον λοιπόν, θέλω να μου πείτε εάν μαζί με τα νέα μέτρα που προτείνονται από πλευρά σας και που εισάγονται, ε, εάν προσπαθείτε να πιέσετε και τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν επιτέλους στη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, μιας πιο αποτελεσματικής δηλαδή διαχείρισης όπως την προτείνετε και εσείς. Και θέλω να μου πείτε εάν κατά, την, ε, κατά τα προγράμματα εξαγοράς ABS θα εξαγοράζονται και οι κλάδοι κινδύνου χωρίς να υπάρχουν κρατικές εγγύησεις ή μόνο εάν υπάρχουν κρατικές εγγύησεις. Και επίσης τα, αναπτυξιακά, τα μοντέλα ανάπτυξη με βάση τα οποία αξιολογήθηκαν τα ABS θετικά μπορείτε να τα δημοσιοποιήσετε γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι. Πρέπει λοιπόν να είναι διαφανές το πόσο σημαντική είναι αυτή η κίνδυνη. Απάντηση. Ευχαριστώ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια εκτίμηση το πόσο, του πόσο μεγάλα ήταν τα κέρδη των τραπεζών Ευχαριστώ, στο LTRO το 2012. Αν υπήρχε όμως κάτι τέτοιο θα σας το διαθέσουμε. Για το δεύτερο σημείο. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου επιτρέπει να διευκρινίσω ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που έχουμε θέσει σε κίνηση. Τα ABS. Θα αγοράσουμε χωρίς εγγύησης τα ανώτερα senior ε, επίπεδα των ABS, senior trenches. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι υπάρχει μια γενική δυσπιστία απέναντι στα ABS που ξεκινάει από τον στρεβλωτικό ρόλο που είχαν αυτά τα ομόλογα κατά τη, για τη δημιουργία, το σχηματισμό μεγάλων ε, οικονομικών κρίσεων. Ωστόσο εδώ πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των ABS εκείνων τα οποία είναι διαφανή, απλά και πραγματικά από εκείνα τα οποία είναι ε, ασαφή και πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν, να τιμολογηθούν. Άρα λοιπόν, εάν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του, ε, της κατάστασης των ΗΠΑ με τα χρεόγραφα που ήταν στηριγμένα στα στεγαστικά δάνεια του 2007 με 20% κίνδυνο ε, αφαιρεγιότητας, την ίδια εποχή ήταν 0,12% στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος αυτός. Με το ίδιο όνομα δηλαδή έχουμε δύο άκρος διαφορετικά είδη χρεογράφων. Τα δικά μας, ABS ήταν απλά, γιατί μπορούσε ο κόσμος να δει τι είδους δάνειο εμπεριέχουν τα ABS, ήταν διαφανή. Και είμαστε σε αυτή την κατηγορία ακριβώς ότι δηλαδή θέλουμε τα ABS ε να προσφέρουν δάνεια στην πραγματική οικονομία. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για τα ABS. Ε μια δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι ότι αγοράζουμε μόνο ένα τμήμα, το senior tranche όπως λέμε από τα ABS, ε το ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή, εάν παρελπίδα τα ABS αποτύχουν, τότε την απώλεια την αναλαμβάνουν πρώτα οι κάτοχοι και του, χρεογράφου και δεύτερον εκείνοι οι οποίοι έχουν το επόμενο επίπεδο, το λεγόμενο μετζάνιν, τον ημιόροφο. Έτσι λοιπόν, εάν φτάσουμε μέχρι τον ημιόροφο, τότε θα χρειαστεί κρατική εγγύηση, αν φτάσουμε στο μετζανίν δηλαδή. Αλλά όταν είμαστε στους ανώτερους ορόφους, στα ανώτερα επίπεδα, δεν χρειάζεται εγγύηση θα χρειαστεί βέβαια και θα δοθεί με βάση τους κανόνες περικρατικών ενισχύσεων, άρα θα πρέπει να είναι και συμβατή αυτή η εγγύηση με την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο τότε θα περάσουμε στον ημιόροφο. Και αν μου επιτρέψετε θα προσθέσω κάτι ακόμη, ότι υπάρχουν πολλά μέτρα που επιτρέπουν αυτά τα EBS να, καταστούν διαφανή. Ένα εκ των οποίων είναι, όπως είπα, το να γνωρίζουμε τι είδους δάνεια εμπεριέχουν, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη και μάλιστα αυτό ήδη έχει προχωρήσει σε μια προσπάθεια ανεξάρτητη πριν από χρόνια, έχει ένα δικό της μητρό ε, καταγραφής αυτών των ABS που θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμο. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρούμε ε, που χρησιμοποιούμε τα ABS είναι ένα σημαντικό κομμάτι των εγγυήσεων που χρησιμοποιούν οι τράπεζές μας για να δανειστούν από την ΕΚΤ. Άρα έχουμε συνηθίσει να διαχειριζόμαστε. Είναι γνωστά τα ABS. Όπως είπα, τα ανώτερα επίπεδα τους κυρίως, Με την υψηλότερη εξοπλιστική προτεραιότητα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας ε, Μάριο Ντράγκη και σας ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Στη διάρκεια της ε, περασμένης νομισματικής περίοδου είχαμε καταγγείλει τα όσα περιλάμβανε το έγγραφο της ΕΚΤΕ σε σχέση με τα TLTRO. Την ε, Παρασκευή πρώιμα επιστράφηκαν 19,9 ε, δισεκατομμύρια των παλαιών TLTRO αλλά κατά τη γνώμη σας είναι σύμπτωση ή, ή μήπως οι τράπεζες χρησιμοποίησαν τα παλαιά TLTRO για να αντικαταστήσουν, να επιστρέψουν ε, μάλλον αυτά. Και έπειτα, εάν δεν επιβάλλουμε υποχρεώσεις, το μόνο το οποίο αναλαμβάνουν είναι τα μπόνους των μάνατζερ και τα χρήματα που γυρνάνε στις τσέπες των ε, χρηματιστών. Αυτοί οι οποίοι άλλαξαν τα TLTRO για ABS δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αντικαθιστούν τον όγκο ε, στην ε, αγορά με το συστημικό κίνδυνο της ε, φούσκας. Δεν γίνεται τίποτα για την πραγματική οικονομία και γι' αυτό και θα παραμείνει χαμηλός ο πληθωρισμός. Πώς πιστεύετε πως θα επιβάλλετε υποχρεώσεις και όχι απλά συστάσεις για τις τράπεζες που παίρνουν χρήματα από το θεσμικό όργανο το οποίο εσείς ε, το οποίο και Έπειτα πώς θα γίνουν πραγματικά χρήσιμα ε, βήματα για τους πολίτες και όχι μόνο για τους φίλους σας της City και του City και του Wall Street, πώς θα απομονώσετε τους ε, ε, κερδοσκόπους γιατί συνεχίζεται το πρόβλημα της φούσκας να υπάρχει. Πώς θα υπάρξουν κάποιες δεσμεύσεις και θα το σκεφτούμε κάπως περισσότερο. Τέλος, τι πιστεύετε για ένα μείγμα κινήτρων νομισματικών και δημοσιονομικών όπως έκαναν η ΕΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου κράχ με επεκτατικές ε, δημοσιονομικές πολιτικές και άφησαν το έλλειμμά τους να αυξάνεται κατά 4 ή 6% κάτω από το ΑΕΠ. Τελικά όμως αυτά απορροφήθηκαν. Μπορούμε να σκεφτούμε μια τέτοια πολιτική για την Ευρωζώνη ή πρέπει να τηλεφωνήσουμε την Γερμανίδα Καγκελάριο για να τη ζητήσουμε την άδεια. Ευχαριστώ. Well, uh, it's a lot of questions. Um, Πολλές ερωτήσεις. Μπορώ να επαναλάβω αυτό που μόλις είπα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, το 80% των πιστώσεων περνά άμεσα από τις τράπεζες. Αυτές είναι οι διαμεσολογητές. Θέλεις λεφτά, πας στην τράπεζα. Είναι μια... κάτι το αναπόφευκτο. Πώς πας στην τράπεζα, Το ένα είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι πιο εύκολες και έπειτα συγκεκριμένα αιτήματα. Ε, αυτή τη φορά δεν έχουμε μόνο συστάσεις γιατί το πρόγραμμα Τέλτρο είναι διαφορετικό από το Έλτρο του 2012 και αυτός ο δανεισμός ρητά στοχεύει την πραγματική οικονομία. Εάν υπήρχαν ε, συγκρίσεις ορόσημα στις ε, διαδοχικές πράξεις, θα, υπήρχε, θα υπάρχουν λοιπόν πράξεις για τα επόμενα δύο χρόνια, όπου οι τράπεζες θα είναι ελεύθερες να δανείζονται στα ειδικά χαμηλά μας, με ειδικά χαμηλά μας επιτόκια, ενώ θα πρέπει να δανείζουν στην πραγματική οικονομία με βάση συγκεκριμένο ορόσημο. Εάν δεν πληρώσουν, ε, δεν δανείσουν μάλλον στην πραγματική οικονομία, θα πρέπει να ξεπληρώσουν όσα δανείστηκαν. Και αυτό ισχύει σίγουρα για τις δύο πρώτες δόσεις ε, και αυτό θα το επαληθεύσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουν τα λεφτά πίσω. Άλλη παρατήρηση. Αντικαθιστούν κάτι από κάτι άλλο, ναι, πιθανότατα. Σημαίνει ότι δεν θα δανείσουν, όχι βέβαια. Θα πρέπει να δανείσουν αργότερα. Δηλαδή είναι μια σημαντική αλλαγή από την προηγούμενη πράξη που είχαμε κάνει, όπως είπα παλαιότερα, όπου είχαμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα χρηματοδότησης να κάνουμε και να αποφύγουμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή στο τραπεζικό σύστημα το 2012. Εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με δανεισμό στην πραγματική οικονομία. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είναι διαφορετικά τα πράγματα και υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει για τι τράπεζε που πρέπει να συμμορφωθούν προ αυτέ. Βέβαια δεν πρέπει να κρίνουμε αυτό το πρόγραμμα μονομένα γιατί θα συνδυαστεί με το πρόγραμμα των ABS και των καλυμμένων ε, ομολόγων. Γι' αυτό διστάζουμε να δούμε μόνο ένα νούμερο γιατί θα είναι το σύνολο και η αλληλεπίδραση αυτών των προγραμμάτων που θα προκύψει προκαλέσουν την αύξηση του μεγέθους του ισοζυγίου μας. Από αυτό θα πρέπει να περιμένουμε κάπως πριν αρχίσουμε να τα κρίνουμε όλα αυτά. Μάλιστα, όταν ε, λαμβάνουμε τις αποφάσεις ε, νομισματικής πολιτικής, πραγματικά δεν σκέφτομαι τους φίλους μου στο City και στο ε, Wall Street. Σκέφτομαι τους Ευρωπαίους πολίτες και σκέφτομαι το στόχο που έχουμε της διατήρησης των σταθερότητας των τιμών, την αύξηση του ποσοστού του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, κάτω από το 2% πάντα, και σκέφτομαι την ανάπτυξη, την απασχόληση, σκέφτομαι κυρίως την ανεργία. Κανένας εδώ δεν έχει στο μυαλό του το City, τη Wall Street. Τώρα, με ρωτήσατε επίσης για το διαχωρισμό ανάμεσα στην τραπεζική δραστηριότητα και τις το εμπόριο ακινήτων. Εδώ οριστικοποιούμε μια γνωμοδότηση που θα δημοσιεύσουμε σύντομα. Και τέλος για την δημοσιονομική πολιτική νομίζω πως έχω καλύψει αρκετά το θέμα ε, και μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο τη σχετική ομιλία μου. Ευχαριστώ. Και τώρα εξ ονόματος των μη γεγραμμένων ο Κέρχοφ Άνεμανς. Θα μιλήσω Ολλανδικά, κύριε Πρόεδρε. Θα θέσω ένα πρόγρα... ένα... μία ερώτηση για το πρόγραμμα IBS, για τους τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίησης. Και τι κάνετε για να κερδίσετε το χαμένο έδαφος από τις στοχευμένες μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης που φαίνεται ότι απέτυχαν. Κατά τη γνώμη μου, Υπάρχει αρκετή ρευστότητα, ε, κυκλοφορεί αρκετό χρήμα. Το πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι το ίδιο το ενιαίο νόμισμα και η έλλειψη διαρθρωτικής ε, εμπιστοσύνης. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ανακεφαλοποίησης ε, των τομέων της οικονομίας, ενώ οι τράπεζες έχουν πολλά λεφτά. Είπατε ότι στο πρόγραμμα αγορών τίτλων προερχόμενος από τυλοποίησεις δεν έχετε τμήματα ενδιάμεσης εξασφάλισης, αλλά μόνο τα τμήματα με άμεση, με τη μεγαλύτερη εξοφλητική προτεραιότητα. Άρα και πάλι οι φορολογούμενοι θα αναλάβουν τον κίνδυνο. Αυτοί θα πληρώσουν τα σπασμένα, όπως και στο παρελθόν. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Νομίζω ότι πραγματικά πήγαμε πάρα πολύ μακριά. Το έχουμε παρατραβήξει το σκηνή και θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο από πού ξεκίνησαν όλα τα πράγματα και από την αρχική κρίση. Τι γίνεται λοιπόν με τους τίτλους αυτούς τελικά. Ποια είναι, τα... Ποια είναι η ρευστότητα που έχετε φανταστεί για τα ABS. Και είναι αλήθεια ότι για να διαχειριστείτε το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσετε ένα αμερικανικό πρότυπο όπως έγινε και στις Ηνωμένε Πολιτείε για την διανομή του βάρους από την κρίση των subprimes. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σημείο, τελείωσα την αρχική μου ομιλία με τη φράση «Η κρίση θα τελειώσει πραγματικά μόνο όταν οι πραγματική οικονομία να κτίσει πλήρω την εμπιστοσύνη τη στην αγορά και την ικανότητα των επιχειρήσεων και την προθυμία του να αναλάβουν κινδύνους, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόληση. Και αυτό θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων. Ε, Ένα από αυτού είναι και η νομισματική πολιτική. Αλλά πιο σημαντικό ακόμα είναι η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων η ενίσχυση της αξιοπιστίας του δημοσιονομικού πλαισίου και η ενίσχυση της διακυβέρνησης ε, της Ευρωζώνης. Πριν από λίγο είπα γιατί πιστεύουμε ότι το είδος των τίτλων προερχόμενων από τυλοποίησης και οι συνιστώσεις ε, των IBS που θα χρησιμοποιήσουμε δεν ε, είναι, ε, είναι επικίνδυνα στοιχεία του ενεργητικού, αλλά εξασφαλισμένα και δεν θα αγοράσουμε μεζανίν τμήμα χωρίς πραγματική δημόσια ε, εγγύηση. Για τον BlackRock δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Δεν ξέρω αν αυτό χρησιμοποιεί, ε, ε, μοίρασε τα subprimes. Εμείς το χρησιμοποιούμε ως σύμβουλο για το σχεδιασμό του προγράμματος. Και η Federal Reserve χρησιμοποίησε τέτοια προγράμματα και τέτοια μέτρα για να σχεδιάσει το δικό της πρόγραμμα πριν από 3-4 χρόνια. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τον BlackRock για να μεταφέρουμε συναλλαγές ή για να αγοράσουμε τα στοιχεία αυτά, τα χρεόγραφα αυτά. Ο ρόλος του BlackRock είναι αμυγός συμβουλευτικός και φυσικά αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και οποιαδήποτε ασυμβίβαστο. Μεριμνούμε ιδιαίτερος για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Τώρα για το δεύτερο γύρο, ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο αντιπρόεδρος Μάρκος Φέμπερ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας συλληπιθώ. Ή αν θα ήταν καλύτερο να ακούσω άλλους ομιλητές. Γιατί πάντα ακούμε την ίδια ιστορία ότι χρειάζεται νέα όθηση στην πραγματική οικονομία, χρειάζεται να διαθέσουμε περισσότερο χρήμα, να πατήσουμε τον γκάζι. Όχι, δεν είμαι πράσινος. Όχι, δεν είμαι πράσινος. Ουδέποτε, ουδέποτε πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, λέτε ότι θα πρέπει να διατηθεί φθηνό χρήμα και νομίζω ότι έχετε δώσει αρκετά κίνητρα, αν κοιτάξουμε το ιστορικό της Κεντρικής Τραπέζας και με το παραπάνω. Βλέπουμε κάποιες αποφάσεις που προτείνονται και οι οποίες έχουν ε, να κάνουν με πρακτική που έχουν υιοθετήσει και άλλες κεντρικές τράπεζες από την Ευρώπη, παραδείγμα της Βρετανίας και οι οποίες προτάσεις σας μιλούν μόνο για πλεονεκτήματα αλλά δεν βλέπω να μιλάτε για παρενέργειες και δευτερεύουσες επιπτώσεις. Ε, έχετε πραγματικά τη βεβαιότητα ότι οι τράπεζες θα συμπεριφερθούν όπως ακριβώς το περιμένετε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος το χρήμα να ε, διαρρεύσει σε άλλους τομείς πέραν της πραγματικής οικονομίας, εκεί δηλαδή που δεν έχει καμία σχέση η οικονομία με τη δημιουργία της συνεργασίας. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να συσχετιστούν και να συνδεθούν αυτά κατά τρόπο πολύ ισχυρό με όρους που θα υποχρεώσουν τις τράπεζες να ακολουθήσουν τις ίδιες αξίες με εμά δεν βλέπω από την άλλη βέβαια πολύ μεγάλη ζήτηση για πιστώσεις. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς η διάθεση κεφαλαίου. Βλέπω ότι δεν έχει εξασφαλιστεί επαρκής ζήτηση από την πραγματική οικονομία για το χρήμα αυτό. Και ξέρω ότι μάλλον θα μπορέσετε να μου δώσετε πιο συγκεκριμένε απαντήσεις, αλλά από πλευρά της ζήτησης υπάρχει δυνατότητα να περιμένουμε ότι θα θεσπιστούν οι κατάλληλες εκείνες δομές, οι πρόσφορες εκείνες δομές, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ροή του χρήματος αυτού προς την πραγματική οικονομία, για να μην περιπέσουμε σε φαύλο κύκλο πάλι. Ο κύριος Δράκη. Είπαμε ότι ενώ συνεχίζουμε αυτήν την ε, νομισματική πολιτική, πράγμα το οποίο θα συνεχίσουμε για αρκετό χρόνο ακόμα, Θέλουμε να έχετε υπόψη ότι η δική μας νομισματική πολιτική με την νομισματική πολιτική άλλων αντίστοιχων αρχών άλλων κρατών, η δική μας νομισματική πολιτική προοδευτικά ε, και όλο και περισσότερο ακολουθεί αποκλίνουσα πορεία. Δηλαδή εμείς ε, παραμένουμε επεκτατικοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα όμως επαγρυπνούμε στο μέγιστο και έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονός ότι αυτό ενέχει και κινδύνους χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Και προφανώς διαρωτώμεθα εάν μέσα στην Ευρωζώνη ήδη διαφέρονται κάποια τέτοια σημάδια κινδύνων. Έχει γίνει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, ανάλυση κατά τη διάρκεια μιας συζητήσεων ε, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών της Βασιλείας πριν από δύο εβδομάδες. Ε, ανάλυση η οποία έδειξε πως η πτητικότητα όντως έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι κίνδυνοι κατά έχουν περιοριστεί σε βαθμό άνευ προηγουμένου και ε, αναπάντοχο θα λέγαμε. Παρόλα αυτά, μέσα στην Ευρωζώνη, ίσως σε άλλες περιοχές να φαίνεται, σε άλλες ε, ζώνες οικονομικές, αλλά στην Ευρωζώνη δεν βλέπουμε την μόχλευση αυτή που θα οδηγούσε σε αύξηση σημαντική στην πιστοτική δραστηριότητα των τραπεζών. Που συνδεδεμένη με τη χαμηλή πτυτικότητα και το χαμηλό κίνδυνο θα μπορούσε να οδηγήσει σε φούσκα. Αυτό λοιπόν δεν το βλέπουμε. Και άμα κοιτάξουμε και συγκεκριμένα κομμάτια, τμήματα της, των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωζώνη, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα σοβαρά μηνύματα υπερβολών. Εάν βλέπαμε κάποια σημάδια υπερβολών, θα ήταν πάντως περιορισμένα τοπικά συγκεκριμένα φαινόμενα και για να τα εντοπίσουμε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μακροοικονομικά μέσα εποπτείας, προληπτικής εποπτείας και όχι γενικευμένα μέσα για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Πράγμα το οποίο όμως όπως είπα δεν διαφαίνεται. Επίσης, υπήρχατε κάποια άλλη ερώτηση. Κύριος Βέμπερ. Ναι, ρώτησα πώς βλέπετε να αναπτύσσετε η πλευρά της ζήτησης για τις πιστώσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχει προσφορά, αλλά ζήτηση δεν βλέπουμε να υπάρχει. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, ζήτηση δεν υπάρχει. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε τις χρηματοοικονομικές εκείνες συνθήκες οι οποίες θα εξασφαλίσουν όταν έρθει η ώρα να εμφανιστεί η ζήτηση, να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε, να την διαχειριστούμε. Είδαμε ταυτόχρονα, για να πούμε και τα θετικά, ότι με τις καλύτερες αυτές ε, συνθήκες χρηματοδότησης βρίσκονται λύσεις μέσα από την πραγματική, φτάνουν δηλαδή αυτές οι συνθήκες στην πραγματική οικονομία. Μην ξεχνάμε τι έγινε μέχρι τα μέσα του 2012, όπου είχαμε τη μία κρίση χρηματοδότησης μετά την άλλη, με επιτόκια πάρα πολύ υψηλά, υπερβολικά υψηλά και αυτό που είδαμε βασικά ήταν ο κατακαιρματισμός του τραπεζικού τομέα στην Ευρωζώνη να οφείλεται στην κρίση του 2012, αλλά να μην έχει ακόμη αντιμετωπιστεί. Να παραμένει δηλαδή ενισχύ. Αυτό λοιπόν θέλουμε να αποτρέψουμε τη ρίζα αυτής της, αυτού του κατακαιρματισμού και όπως είπα η νομισματική πολιτική προϋποθέσεις γεννά αλλά τον κύριο και τον κυρίαρχο ρόλο θα για την ανάπτυξη, για, τη, τα κίνητρα, για τη ζήτηση θα τον έχουν α, οικονομικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είπατε ότι θέλετε να δώσετε κίνητρα στις τράπεζες. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Το 2010 ως ε, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας ε, στείλατε ένα τέτοιο μήνυμα στις Ιταλικές τράπεζες λέγοντάς τους να κόψουν τα επιτόκια. Τώρα, ενώ η ΕΚΤ θα είναι επόπτης των εθνικών τραπεζών, δεν ε, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν ε, επέβαλε πάγωμα των ε, τοκομεριδίων. Γιατί δεν το κάνατε αυτό, γιατί δεν προσπαθήσατε να επιβάλλετε πάγωμα των τοκομεριδίων και ρωτώ στο συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικά περιορισμένων προσπαθειών των τραπεζών αυτή τη στιγμή για να αντλήσουν φρέσκο κεφάλαιο πριν από τα ε, δοκιμές αντοχής. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη, αν και μάλλον θα είναι βαρετή για σας, αλλά θέλω να επανέλθω στα ABS. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι περί πρόκειται. Βασικά, Εάν ε, η ομάδα ABS που αγοράζεται δεν περιέχει κίνδυνο, δεν καταλαβαίνω σε τι θα βοηθήσει την δίωδο της πίστοσης. Και έπειτα, επειδή είναι σχετικά περιορισμένο κομμάτι, πώς μπορεί να φτάσει σε όγκους που μπορεί να επηρεάσουν άλλες διόδους, όπως το, η διόδος των ισοτιμιών. Πώς λοιπόν θα λειτουργήσουν όλα αυτά, ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Για το πρώτο σας ερώτημα, οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ δεν είναι οι αρμοδιότητες υποπτικές στην φάση αυτή. Όταν η ΕΚΤ θα αναλάβει πλήρως τις εποπτικές της αρμοδιότητες, θα είναι σε θέση να ζητήσει περιορισμούς στα τοκομερίδια, περιορισμούς στους μισθούς, όπως το έκανα τότε. Έχετε δίκιο στην Banca d'Italia και να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη για να ε, ενισχύσουν την κεφαλαϊκή βάση. Για την ώρα δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τους εθνικούς υπόπτες. Και μάλιστα ορισμένοι το έκαναν αυτό που λέτε. Ενώ άλλοι όχι. Εξαρτάται από την κατάσταση σε κάθε χώρα. Δεύτερη σας ερώτηση τώρα. Μιλήσατε για δύο σημεία. Το πρώτο είναι πώς μπορεί η αγορά μόνο μεγάλων ομάδων μέχρι ότου να δώσει κάποια χώρα ή κάποια τράπεζα μια εγγύηση, πώς μπορεί να ελευθερώσει χώρο στο ισοζύγιο της τράπεζας. Αυτό εν μέρει αληθεύει, αλλά δεν όχι απόλυτα το κεφαλαικό βάρος στο λιγότερο επικίνδυνο τμήμα είναι πολύ χαμηλότερο από ότι στις, ε, πιο στα πιο επικίνδυνα τμήματα δεν είναι μηδενικό, οπότε σε κάποιο βαθμό επηρεάζει την πτυχή του κεφαλαίου. Από την πλευρά της χρηματοδότηση βεβαίω πληρώνει την επίπτωση τέλτρο. Όσον αφορά το μέγεθος, το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της αγοράς. Δεν είναι σαφές ακριβώς ποιο θα είναι το μέγεθος της αγοράς που θα αντιμετωπίσουμε, διότι αν δούμε τα πράγματα με την ε, εικονική τους αξία. Έχουμε αρκετά μεγάλη αγορά, αλλά μετά αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε μια σειρά ABS που δεν ανταποκρίνονται στις προαπαιτήσεις μας, διότι θέλουμε να είναι απλά, να είναι διαφανή, να περιλαμβάνουν ε, δανεισμό στην πραγματική οικονομία και ούτω καθεξής. Έπειτα λοιπόν αυτό το μειώνουμε και λέμε πόσο από αυτό το κομμάτι που είναι ακόμα μεγάλο ανήκει στη δευτερεύουσα αγορά και πόσο έχουν στην κατοχή τους οι επενδυτές. Ένα μεγάλο τμήμα όλων αυτών το έχουν οι επενδυτές. Οπότε εμεί θέλουμε να μπούμε σε αυτή την αγορά, να διευρύνουμε τη δευτερεύουσα αγορά και να επίσουμε τους επενδυτές να εμπορευθούν τα κομμάτια που έχουν στην κατοχή τους, γιατί πιστεύουμε ότι το μέγεθος αυτής της αγοράς είναι ενδογενές, δηλαδή ανταποκρίνεται στο δικό μας ρόλο και στις ε, πρωτοβουλίες μας. Τέλος, διερωτάστε ποιες είναι οι επιπτώσεις στις συναλλαγματικές οτιμίες, Όπως γνωρίζετε, οποιοδήποτε σχόλιο για τις ισοτιμίες είναι πολύ λεπτό, γιατί έχουμε δεσμευτεί στη G20 να χειριζόμαστε τις ισοτιμίες ως ένα θέμα κοινού συμφέροντος. Και έχω πει επανειλημμένως ότι η ισοτιμία δεν είναι στόχος πολιτικής, αλλά είναι σημαντικό στοιχείο για τη σταθερότητα των τιμών και την ανάπτυξη. Είδαμε την αποδυνάμωση των, ε, της συναλλαγματικής ισοτιμίας τις τελευταίους έξι μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλα Μασούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του G20. Εδώ και έξι χρόνια υπάρχει το G20. Δημιουργήθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Μπορείτε να μας πείτε συντομία που χάρη στις προσπάθειες του G20 η διεθνής κοινότητα γενικώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικώ ε, σημείωσαν σημαντική πρόοδο και σε ποια σημεία έχουμε μείνει πίσω. Είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι σήμερα για να προλάβουμε ή να αποτρέψουμε στιμικό κίνδυνο ε, όπως αυτός ε, του 2008 και ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι σύμπτωση που θέτει το ερώτημα σε κάποιον που δεν είχε παραστεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του G20. Πάντως, στις τελευταία συνεδριάσεις του G20 δόθηκε έμφαση στην ολοκλήρωση της ε, χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας, μια προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές του 2008. συζητήθηκε και μάλιστα εκτενώς ε, το θέμα της αποκατάστασης της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, αυτό το θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα στο G20. Θα έλεγα ότι το G20 ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα ε, ομάδα για την προώθηση της, ε, της προόδου στην, ε, στις νέες χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις. Προκειμένου οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι τράπεζες να γίνουν πιο ανθεκτικές σε κρίσεις που πάντα είναι πιθανό να συμβούν. Είχαμε μεγάλη πρόοδο στο σχεδιασμό, αλλά πολύ πιο περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή. Με την αποκατάσταση εμπιστοσύνης χρηματοπιστωτικές αγορές, μία αίσθηση κατεπήγοντος, ώστε και οι εποπτικές αρχές να συνεργαστούν προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κανονισμό, αυτή η βούληση έχει μειωθεί. Η βούληση για συνεργασία. Αυτή ήταν η βασική συμβολή του G20 και χαίρομαι που η ομάδα αυτή συνεχίζει τη συζήτηση για τα θέματα αυτά και ζητά την πραγματοποίηση περισσότερη πρόοδου. Ένα άλλο θέμα που στήθηκε στην Αυστραλία ήταν η ανάπτυξη, οι σωστές οικονομικές πολιτικές που τονώνουν την ανάπτυξη και ένα συναφές θέμα, το θέμα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των διαφόρων ζωνών αλλά και του, τους κινδύνους μετάδοσης των δικών μας πολιτικών σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό το θέμα έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στις διαδοχικές συζητήσεις του G20. Ευχαριστώ. Αλέσια Μούσκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Εγώ θα επανέλθω στι ανησυχίε που ανέφεραν πολλοί σήμερα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των νομισματικών πολιτικών που ασκούνται και τον αντίκτυπο που έχουν αυτέ επί της ε, πραγματικής οικονομίας αλλά και ε, σε σχέση με την ανάγκη πιο στεναρού συντονισμού ανάμεσα στι νομισματικέ πολιτικέ, στις ε, διευθυντικές μεταρρυθμίσει των χωρών και μια ερώτηση όσον αφορά την ολοκληρωμένη ζήτηση. Κατά τη γνώμη μου βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της ευρωπαϊκής πολιτικής με ένα σχέδιο για τις δημόσιες επενδύσεις που έχει ανακοινωθεί και που θα δοθούν λεπτομέρειες τις επόμενες εβδομάδες και διερωτώ με και σας ρωτώ κατά τη γνώμη σας ποιες μπορούν να είναι οι προτεραιότητες για αυτές τις επενδύσεις έτσι ώστε να υπάρξουν να μην υπάρξουν πολλές ε, επιβραδύνσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και κατά δεύτερο λόγο στην ομιλία σας στην Jackson Hall που ακούσαμε και στο Μιλάνο μείνατε, επιμείνατε στην ε, στο, στην αρνητική επιρροή της ανεργίας στις νομισματικές πολιτικές και γι' αυτό και αναφέρομαι στην, ε, υπό το φως μάλλον των ισνών αποτελεσμάτων που είχαν οι δράσεις ε, κατά της ανεργίας. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξει η προσέγγιση και τι ιδέα έχετε για αυτή την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Ασφάλισης κατά της ανεργίας με πολύ διαφορετική προσέγγιση γιατί θα επηρεάσει και τις εθνικές ασυμμετρίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις σας είναι ευρύτατες και σε κάποιο βαθμό εκτός ε, ε, θέματος. Σίγουρα όμως ένα από τα θύματα της κρίσης ήταν οι επενδύσεις. Ε, οι ιδιωτικέ και οι δημόσιες. Εν γέννη οι επενδύσεις σήμερα βρίσκονται σε ένα επίπεδο νομίζω σε σχέση με το ΑΕΠ είναι σε ένα επίπεδο που δεν έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Οι δημόσιες επενδύσεις έχουν γίνει επίσης πολύ χαμηλά, έχουν πέσει πολύ χαμηλά για τον απλό λόγο ότι όταν ε, οι χώρες πρέπει να εξηγιάνουν τη δημοσιονομική τους πολιτική και τους προπολογισμούς τους κάνουν το πλούστερο και το ευκολότερο που μπορούν να κάνουν ε, βιαστικά βιαστικά σε επίγουσα δηλαδή κατάσταση δηλαδή να αυξήσουν τους φόρους και να περικόψουν τις επενδύσεις. Αυτά όλα συνδυασμένα σε μια φάση κρίσης ε, απώλειας εμπιστοσύνης ε, δημιουργούν μια πολύ σοβαρή κατάσταση για την ενέργεια και κατά κάποιο τρόπο Αυτή είναι και η κυκλική συνιστόσα της ανεργίας στην Ευρωζώνη. Λέμε ότι είναι διορθωτικό το θέμα, ότι έχουμε σοβαρές, σοβαρά εμπόδια για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωζώνη και είναι και αλήθεια αυτό σε μεγάλο βαθμό. Αλλά επίσης είναι μια κυκλική συνιστόσα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί Η επιστροφή λοιπόν στις επενδύσεις είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό πολύ συχνά μιλώ για φιλική προς την ανάπτυξη ε, δημοσιονομική εξυγίανση και αυτή η επιστροφή στις επενδύσεις θα πρέπει ωστόσο να συμβαδίσει με δράσεις οι οποίες στόχο θα έχουν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα στις προοπτικές αυτής της οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο Μπέρντ Λάγκερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια, με τη σαφή σας εκείνη δήλωση από το Λονδίνο, μπορέσατε να αποτρέψετε από τη μια μέρα στην άλλη την κερδοσκοπία βάρος κρατών. Πολύ καλά κάνατε. Δεν θέλω λοιπόν να διατυπώσω για το M1 ή για το M3 ερωτήσεις. Ε, πρόκειται για δείκτες ως προς την ε, απουσία εμπιστοσύνης ή την παρουσία συγκυριών. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο για το πώς κρίνεται δηλαδή την νομισματική πολιτική Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωζώνης. Έχετε εσείς ή σκοπεύετε να, περι... να μειώσετε ακόμη περισσότερα τα επιτόκια. Έχετε όπως η Federal Reserve την πρόθεση για εξαγορές, ε, να διαθέσετε χρήμα μάλλον στην αγορά. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν βραχυπρόθεσμα σημαντικές διαταραχές στην αγορά. Και δεύτερον, η ΕΚΤ βλέπει μία δυνατότητα αυτή τη χαλαρή νομισματική πολιτική να την ε, κλείσει, να την ε, αλλάξει πριν το 2016 και όχι μετά το 2016 όπως είπατε εσείς. Και τρίτον, βλέπουμε ότι έχει πέσει το ευρώ σε σχέση με το δολάριο δεν έχει φτάσει βέβαια στην πλήρη ισοτιμία, αλλά πιστεύετε ότι με χαμηλό επιτόκιο μπορεί να αποτρέψετε τον κίνδυνο οι επενδυτές να προτιμούν το δολάριο. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε μια σαφέστερη εικόνα για το τι φοβάστε, τι ελπίζετε και πώς κρίνετε την κατάσταση. Κύριε Δράκη, ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. όταν διάφορες ζώνες του κόσμου και ιδιαίτερα μεγάλες όπως οι ΗΠΑ ή η Ευρωζώνη ακολουθούν αποκλίνουσες πορείες στην νομισματική πολιτική πρέπει, οφείλουμε και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού μάλιστα να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις κινήσεις ο ένας του άλλου και να υπάρχει επικοινωνία ή τουλάχιστον να φροντίζουμε ή επικοινωνιακή πολιτική καλύτερα των αποφάσεών μας να μην οδηγεί σε απρόβλεπτες ή αθέλητες διαταραχές και κινήσεις στις αγορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προβλήματα. Και ακριβώς αυτό κάναμε πριν από λίγο, αυτό το είδαμε πριν από λίγο καιρό γιατί υπήρξαν κάποιες τρευλώσεις συνθήκες αγοράς. Τόσο λοιπόν εμείς με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και ε, ομόλογοι μα ανά τον κόσμο γνωρίζουν πολύ καλά ότι τέτοιου είδου αποφάσει πρέπει να λαμβάνονται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να ανακοινώνονται, να κοινοποιούνται με όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή επίση. Πρόθεσή μα φυσικά, πρόθεση είναι εν γέννη να αποτρέπεται κάθε ε, απρόσμενη, αθέλητη, ανεπιθύμητη στρέβλωση και ταραχή, διαταραχή στι αγορέ. Πράγμα το οποίο πιστεύω μέχρι τώρα έχουμε επιτύχει. Για τη δεύτερη σας ερώτηση πότε θα σταματήσουμε αυτή την χαλαρή νομισματική πολιτική. Θα τη σταματήσουμε όταν θα έχουμε εκπληρώσει την εντολή μας, που είναι δηλαδή να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα του πληθωρισμού στο 2%. Κοντά στο 2%, κάτω από το 2%. Αυτή είναι η πρωταρχική, αυτός είναι ο πρωταρχικός, αν όχι ο μόνος στόχος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και πάντως είναι ο κύριος στόχος μας όπως καταγράφει η συνθήκη. Για τις προβολές και προβλέψεις. Προς το παρόν, η νομισματική πολιτική μας παραμένει χάλαρη και όπως είπα στο βαθμό που χρειάζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ήδη συζήτησα το θέμα των πιθανών παρεπόμενων συνεπειών ε, αυτής της πολιτικής. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα, αλλά όπως είπα παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και τη διάσταση αυτή. Δεν ε, εφησυχάζουμε. Για την τρίτη σας ερώτηση και την ισοτιμία που όπως είπα είναι πολύ δύσκολο διοικητής κεντρικής τράπεζας τόσο μεγάλης να κάνει σχόλια για ισοτιμίες. Έχουμε όλοι συλλογικά στο G7 και στο G20 στις δηλώσεις για τις ισοτιμίες που κρίνουμε ως ζήτημα κοινού συμφέροντο, έχουμε επιλέξει μια πολύ προσεκτική γλώσσα όλοι. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα να τοποθετηθώ. Αλλά επανερχόμενο και παρατρέποντα την πρώτη σα ερώτηση, παραλαμβάνω ότι έχουμε νομισματικέ πολιτικέ σε αποκλίνουσα πορεία και θα παραμείνουν σε αποκλίνουσα πορεία καθώς προχωρά η ανάκαμψη στις ΗΠΑ και ενισχύεται ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ προς τους στόχους τους ενώ σε εμά τα πράγματα βαίνουν πιο βραδέως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Όλε Λούτβιξον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και χαίρομαι που σας βλέπω κύριε Δράγκη. Πρόσφατα ο αντίκτυπος της ανεργίας ελήφθη υπόψη κάπως στην νομισματική πολιτική. Η ανεργία ο σημαντικός παράγοντας θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη γνώμη μου. Γιατί η ανεργία στην Ευρωζώνη είναι υψηλή και ειδικά η διαρθρωτική ανεργία πολύ υψηλή. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να πετύχουμε το στόχο του πληθωρισμού γύρω ή κάτω από το 2% με τόσο υψηλή ενεργεία. Θεωρείτε ότι θα υλοποιήσετε το στόχο σας ή θεωρείτε ότι πρώτα θα πρέπει να μειωθεί η ανεργία αισθητά και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο ώστε να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υλοποιήσει το στόχο του πληθωρισμού του 2%. Γιατί η ανεργία επηρεάζει και τους μισθούς που και αυτοί έχουν πάρει μια πτωτική πορεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δράγκη. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την αδιεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής. Και η ερώτηση αποδέχεται τουλάχιστον δύο απαντήσεις που είναι και συμπληρωματικές μεταξύ τους. Το 2011 ο πληθωρισμός ήταν 3%. Τώρα είναι 0,4%. Διαρωτηθήκαμε λοιπόν. Πού οφείλεται αυτή η μείωση στον πληθωρισμό. Σίγουρα, δύο τρίτα της μείωσης αυτής για το πρώτο χρονικό διάστημα μεταξύ του 2011 και των τελών του 2012 η πτώση οφειλόταν στο διάστημα αυτό στην ε, μείωση, στη μείωση της τιμής του πετρελαίου και στη μείωση των τιμών των τροφίμων. Υπήρχε και ένας τρίτος παράγοντας, ένας τρίτος λόγος που εμφανίστηκε όμως αργότερα στα τέλη του 2012 και στις αρχές του 2013 και ήταν το γεγονός ότι σε πολλές χώρες και σε όλες τις χώρες με προγράμματα διάσωσης είχαμε μια σχετική προσαρμογή των τιμών και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας που απαιτούσε μείωση των τιμών που για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό φυσικά συνέβαλε στη μείωση του ποσοστού του πληθωρισμού. Στη συνέχεια η μείωση αυτή, παρόλο που σε τιμή δολαρίου ε, οι τιμές των τροφίμων και οι τιμές του πετρελαίου δεν μειώθηκαν περαιτέρω, σε εμά ε, είχαμε ε, και ένα ευνοϊκό ποσοστό συναλλαγματικής ισοτιμίας που συνέβαλε και αυτό, η συναλλαγματική ισοτιμία σχέση με το δολάριο συνέβαλε στη μείωση του πληθωρισμού, στη μείωση του τιμάριθμου. Εν τω μεταξύ βέβαια η ανεργία εκτοξεύθηκε στα ύψη στην Ευρωζώνη συνολικά. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ανεργία και η χαμηλή ζήτηση που συνοδεύει την υψηλή ενέργεια, συμβάλλουν στην παραμονή του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα, στη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα. Πολύ συχνά με ρωτάτε πώς υπερτιμήσατε και γιατί υπερτιμήσατε τα μοντέλα σας, γιατί υπερτίμησαν τον πληθωρισμό επανειλημμένος. Ο λόγος είναι ότι όλα αυτά τα μοντέλα στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένες εικασίες για τις ε, τεκμήρια για, τις, ε, για τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις τιμές πετρελαίου και τροφίμων. Οπότε οι προβλέψεις για τις τιμές αυτές ήταν εσφαλμένες με αποτέλεσμα να κάνουμε υπερτίμηση του πληθωρισμού. Και μέχρι πρόσφατα θα λέγαμε ότι αυτά τα λάθη στις προβλέψεις οφειλόταν κυρίως ε, σε λάθη στις δικές μας πιθανολογίες εικασίας. Πάντως ένα ποσοστό 20% των λαθών μας οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Ένα πέμπτο των λαθών μας οφείλεται, για παράδειγμα, στην ανεργία. Και συμφωνώ μαζί σας ότι η ανεργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση χαμηλού ποσοστού πληθωρισμού. Ευχαριστώ. Ράιαν Χάιας. Ευχαριστώ πολύ. Και καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Ντράγκη στην Επιτροπή μας. Η πρώτη ερώτηση. Θα είναι να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις για, το, ε- για τα ABS ε και τη χρησιμότητά του για τις τράπεζες. Είπατε ότι είναι 80% του συνόλου του δανεισμού σε όλο το σύστημα για τις τράπεζες βέβαια και εκείνες οι οποίες έχουν περάσει από τα τεστ αντοχής και δείχνουν καλή κεφαλαιοποίηση. Και το ρωτάω αυτό για το εξή λόγο. Αυτή η χρηματοδότηση του ημιορόφου του Μετζανίν μπορεί να διαγνώσει, μπορεί να καταγράψει και ενυπόθηκα δάνεια, τα λεγόμενα tracker mortgages, μέσα στο Μετζανίν, στη χρηματοδότηση Μετζανίν. Και δεύτερον, από την προηγούμενη μας συνάντηση στο Στρασβούργο. Θα είδατε φαντάζομαι απόφαση του Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, της Δημοκρατίας Ιρλανδίας, να γίνει ε, έρευνα σε σχέση με το ζήτημα των εγγύσεων στις τράπεζες και την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα στην Ιρλανδία. Θα, ζητήσει, θα καλέσει μάρτυρες, πολιτικούς, ε, ε, τραπεζίτες και βέβαια και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν σε μια τέτοια δημόσια έρευνα του Κοινοβουλίου μας πώς μπορεί να συμβάλλει και αυτό το λέω δεδομένου ότι ο προκατοχός σας κύριος Τρισέ είχε αρνηθεί να συνεργαστεί και να έρθει να καταθέσει ως μάρτυρα σε αυτή την έρευνα. Η οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Και είχε δηλώσει ο κύριος Τρισέ ε, ότι δεν σκοπεύει να το πράξει. Θέλω λοιπόν να μου να κάνετε και κάποια κρίση σε σχέση με αυτή τη δήλωσή του, την εποχή που, είχε, που κατήχε δημόσιο αξίωμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν τι θα πράξει, πώς μπορεί να διευκολύνει την ε, έρευνα αυτή, την, την Εκθεστική Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας όταν ξεκινήσει. Απάντηση. Ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτηση, δεν ξέρω αν θα περιλάβουμε τα tracker mortgages. Θα σας δώσω μια απάντηση σε μεταγενέστερο στάδιο τα ABS που θα αγοράσουμε έχουν βέβαια ε, εγγύη ε, δάνεια με ομόλογα από αποστεγαστικά δάνεια. Το θέμα όμως είναι, και αυτό πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, κινδυνεύουμε να τροφοδοτήσουμε μία φούσκα αν το κάνουμε αυτό. Η απάντηση είναι μάλλον όχι, διότι υπάρχει ένα περιθώριο από την αγορά αυτών, την εξαγορά αυτών των στεγαστικών ε, ABS. Υπάρχει ένα περιθώριο όμως στους ε, ισολογισμούς των τραπεζών. Δεν καλύπτεται αυτομάτως ο χώρος αυτός και άρα δεν φουσκώνει η αγορά. Πάντως θα προσέξουμε πάρα πολύ. Για τη δεύτερη ερώτηση και παρατήρηση. Δεν έχω να σας δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Θα το μελετήσουμε προσεκτικά. Θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Δεν είχαμε την ευκαιρία ακόμα να το συζητήσουμε. Κύριο Σέις, συμπληρωματικά, εσείς όμως πώς κρίνετε την ε, δήλωση του κυρίου Τρισέ ότι δεν σκοπεύει να έρθει σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Ενώ κατήχε δημόσιο αξίωμα και λάμβανε αποφάσεις ως εκ του αξιώματός του εκείνη την εποχή. Πώς το κρίνετε αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι δική μου η άποψη, δεν είναι η άποψη του Μάριου, είναι η άποψη του, κεντρικού, του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Μόνο με βάση αυτό μπορώ να σας απαντήσω. Φαντάζομαι στην προσεχή συνεδρίαση που θα έρθω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαΐ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Τράγκη, Πολύ σύντομα ε, παραπέμπω και πάλι στην ομιλία σας στο Jackson Hole όπου μιλήσατε για την υποστήριξη της ε, πολιτικής της ζήτησης και της αγοράς για την Ευρωζώνη και την Ευρώπη στο συνολό Τη Βλέπουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και την προσαρμογή των επιχειρήσεων ως προς την ε, προσφορά. Για τη ζήτηση όμως, όταν λέτε α, βελτίωση τη ζήτηση σε ποιον απευθύνεστε, ποιον έχετε υπόψη, τι είδους περιθώριο βλέπετε, υπάρχει δυνατή, δηλαδή δυνατότητα να γίνει διαπραγμάτευση αυξήσεων των μισθών, ώστε να βελτιωθούν οι μισθοί σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να ενισχυθεί η εσωτερική κατανάλωση ώστε να βελτιωθώ η κατάσταση με τις μικρές εντάξεις. Μπορείτε να δώσετε κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις, ενδεχομένω και για κάθε χώρα της Ένωσης. Και δεύτερη ερώτηση, για να επανέλθω στην ερώτηση της συναδέλφου Μόσκα για το δημόσιο χρέος. Είπατε ότι τα περισσότερα κράτη ενισχύουν τους φόρους τους και περιορίζουν τις δημόσιες επενδύσεις τους. Συμμερίζομαι αυτή την επίκριση. Βέβαια πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με τους στατιστικούς κανόνες της Ευρώπης, δηλαδή την υποχρέωση να ακολουθούν τις εστάσεις της Eurostat και τις επιλογές της Eurostat, γιατί αν παρακολουθήσουμε πιο προσεκτικά, τίποτε δεν καταγράφεται από το, από το ενεργητικό των κρατών ε, και το συλλογικό, τον συλλογικό πλούτο των τοπικών και περιφερειακών αρχών γιατί για την πατρίδα μου το Βέλγιο θα είχαμε 50% επενδύσεων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για, όλη, για όλο το Βέλγιο και 7% του συνολικού δημοσίου χρέους. Άρα και αν θέλουμε τα 300 δισεκατομμύρια των ευρώ για τις επενδύσεις, τουλάχιστον όσον αφορά το δημόσιο τομέα, να αποδώσουν, δεν θα έπρεπε να υπολογίζουμε και τις παραγωγικές επενδύσεις για τις τοπικές περιφερειακές αρχές, την χρηματοδότηση και από τις κρατικές αρχές ενδεχομένως βιομηχανικών ζωνών και άλλες μεγάλες επενδύσεις παραγωγικές ως περιορισμό του χρέους. Και ένα άλλο τεχνικό μάλλον ζήτημα που έχει να κάνει της, ε, την υποχρέωση για μπέιλιν των ε, προνομιούχων ε, πιστώσεων, δανειστών, τι μπορεί να γίνει ως προς τον κίνδυνο του κατακαιρματισμού εάν το πεδίο αυτού του Μπέιλινγκ είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα πιο ευάλωτα κράτη. Δεν θα αποτελεί αυτό κίνδυνο για το μέλλον. Oh, uh, Απάντηση. Όντως, όντως, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, ε, της αποκατάστασης του πληθωρισμού η νομισματική πολιτική ώστε να επανέλθει στο 2% κάτω από το 2%. Στην τέτοια κατάσταση λοιπόν η ίδια νομισματική πολιτική δεν επαρκεί. Θα χρειαστούν και άλλες πολιτικές. Και υπενήχθην το, γεγονός αυτό και την κρίση αυτή και στον λόγο στον οποίο αναφερθήκατε κι εσείς. Άρα θα πρέπει να δώσουμε νέες προτεραιότητες στους προπολογισμού ε, και να δώσουμε περισσότερες επένδυσεις, να ενισχύσουμε τις ενισχύσεις. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των κρατών που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο και εκείνων που δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο. Όπως είπα και νωρίτερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συστήσει στις ειδικέ ε, συστάσεις ανακράτος, έχει όντως συστήσει τέτοιου είδους πολιτικές. Για δε τις χώρες που δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο, θα πρέπει αυτές να αναδιαρθρώσουν τις ε, ε, προτεραιότητες τους ως προς την διάρθρωση των προϋπολογισμών τους προκειμένου να ενισχύσουν τις παραγωγικές επενδύσεις ταυτόχρονα όμως περικόπτοντας τις μη παραγωγικές δαπάνες για το Μπέιλιν. Από το 2016 και μετά, αν δεν απατώμε. Μήπως ήταν και 15 ή 16. Έχουμε το BRRD, ε, την, οδηγία δηλαδή για την ε, αποκατάσταση για την ανάκαψη και εξυγίαση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ε, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή και θα φέρει τα αποτελέσματά της. Νομίζω ότι οι αγορές και οι τράπεζες ήδη αποδέχονται αυτή την εξέλιξη με αρκετή αισιοδοξία, με μια ε, φυσιολογική και ψύχρεμη θα έλεγα αντίδραση, δεν προκύπτει δηλαδή πανικό στις αγορές λόγω αυτών των νέων κανόνων που αρχίζουν να ισχύουν. Ευχαριστώ. Τελευταίος μας ο ο κύριος Γεώργιος Χρήστος. Κύρτσο, συγγνώμη. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντράγκη που είναι μαζί μας και έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα και η άλλη είναι ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται πω η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα νέο δανειακό πακέτο από τους επιστοτές της Ευρωζώνης και ότι η χώρα είναι έτοιμη να ακολουθήσει το δρόμο της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και να καλύψει τις οικονομικές τη ανάγκες στις διεθνεί αγορές. Έχω την εντύπωση κύριε Ντράγκη, διαβάζοντα τον τύπο, ότι θα προτιμούσατε ένα νέο πακέτο στήριξης ε, που θα συνοδευόταν από τον αυστηρό έλεγχο της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και ότι απαιτείται περισσότερες εγγυήσει από την ελληνική πλευρά για να βοηθήσετε τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ώστε να παρέξει περισσότερη ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Και τώρα, η είναι αλήθεια αυτό ή όχι, και η ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ερώτηση. Τώρα, σε σχέση με το αύξηση του ποσοστού του πληθωρισμού, στο 2 περίπου της 100 δεν συνδέεται με άλλους βασικούς στόχους ε, που έχετε θέσει για να δεχτούμε την πολιτική και την οικονομική τριβή στο μέλλον που θα μπορούσε να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που μόλις μας περιγράψατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω μια φορά ακόμα ότι στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες δεν υπάρχει παζάρι. Δεν γίνεται διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την κυβέρνηση. Εμείς ακολουθούμε την εντολή μας και οι κυβερνήσεις ακολουθούν τη δική τους εντολή. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να, μάλλον συχνά προκύπτει ε, αυτή η κατάσταση. Μας έχουν πει δηλαδή ότι μειώνουμε τα κίνητρα για τις κυβερνήσεις ώστε να μεταρρυθμιστούν, να προβούν σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα αυτό το επιχείρημα ε, αφήνει απ' έξω το εξή, ότι εμείς έχουμε μια εντολή και ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι υποκατάστατο των διαφορετικών ε, μεταρρυθμίσεων. Άρα εξαρτάται από τις κυβερνήσεις και ειλικρινά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι κάποιες κυβερνήσεις αντιδρούν σε κίνητρα επιτοκίων, ας πούμε αν μειωθούν τα επιτόκια δεν μεταρρυθμίζονται και δεν αντιδρούν στα εκατομμύρια ενέργων που έχουν στη χώρα τους. Αυτό θα έπρεπε να είναι πιο, πολύ πιο ισχυρός ε, παράγοντας που να οθήσει τις κυβερνήσεις να προβούν σε διαφορετικέ αλλαγές ε, μεταρρυθμίσεις από ότι ένα, μια ποσοστιαία μονάδα πάνω ή κάτω στα επιτόκια. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να αναμειχθούμε. Έπειτα ε, η ΕΚΤ αναγνωρίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο την οποία έχει σημειώσει η Ελλάδα όσον αφορά την λήψη διαφόρων ε, δημοσιονομικών μέτρων στον προπολογισμό, στις διαφορετικές αλλαγές ε, και βεβαίως όχι μόνο η ΕΚΤ αλλά και οι αγορές το έχουν σημειώσει αυτό και προσέφεραν στην Ελλάδα ε, έκτακτες, ε, έκτακτους όρους χρηματοδότησης που βασίζονται στην προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων και ότι θα προβεί σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από το τρέχον πρόγραμμα. Σκεφτόμενοι μάλιστα πως η τρέχουσα κατάσταση στις αγορές θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη, θα πρότεινα όλοι μας να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη χρονική στιγμή ώστε να συνεχίσουμε στην προσπάθεια μεταρρύθμισης χωρίς να οδηγηθούμε σε βαρέσκεια. Και έπειτα, για το κατά πόσο υπάρχουν τριβές ή όχι. Ε, κοιτάξτε, κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι υπάρχουν και ε, διαπραγματεύσεις. Όχι, οι τριβές υπάρχουν διότι έχουμε συγκεκριμένη εντολή και οι κυβερνήσεις δική τους εντολή διαφορετική και εμείς ε, αυτή την εντολή θέλουμε να εφαρμόσουμε και επιμένουμε σε αυτή και να σας διαβάσω μόνο ένα κομμάτι της δήλωσης που έκανα στην αρχή. Με τα προγράμματα αγορών ξεκινάμε μια μετάβαση από, μια, από ένα πλαίσιο νομισματικής πολιτικής που βασικά εδραζόταν σε παθητικές ε, πολιτικές, σε πιο δραστήρια διαχείριση του ισοζυγίου μας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ντράγκη. Νομίζω πως ε, ήταν πολύ καρποφόρος ο διάλογός μας. Ο επόμενος νομισματικός διάλογος θα είναι στις 17 Νοεμβρίου και νομίζω μπορούμε να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τον Πρόεδρο Ντράγκη για την παρουσία του και προσβλέπουμε στην επόμενή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Please. Let me first. Uh, Θα ήθελα να καλωσορίσω ολόθερμα τον Επίτροπο Μπαρνιέ που έχει την καλοσύνη να έρθει για την ανταλλαγή απόψεων και να αποτίσω φόρο τιμής στο έργο του και στη στράτευσή του προκειμένου να γίνει πιο αθεκτικός ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός κλάδος και να καταφέρουμε να δώσουμε σάρκα και οστά στην Τραπεζική Ένωση. Και μάλιστα ο προκατοχός μου, της, ο πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ εργάστηκε και συνεργάστηκε πολύ στενά μαζί σας και είναι σημαντικό σε αυτή την τελευταία μας συνάντηση να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το έργο σας, τη συμβολή σας και την αγαστή συνεργασία που είχαμε ανέκαθεν. As, as announced... Η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ήθελε κάποιες εξηγήσεις για τις κατεξουσιοδότησης για τις και τα εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για την ανάκαμψη και Εξηγίαση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης καθώς και τη συνεισφορά στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Επίσης θα θέλαμε να εξετάσουμε και να συζητήσουμε άλλες σημαντικές κατεξοδότηση πράξεις που αναμένεται να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ρευστότητα, τη μόχλευση και τη συμπλήρωση της φαρενκιότητας 2. Και χαιρόμαστε που ήρθατε εδώ για την πρώτη αυτή εξέταση των καταξιδότηση και των πράξεων και το σχετικό έλεγχο, αλλά φαντάζομαι θα επεκταθείτε και σε άλλα σημεία στην ομιλία σας. Πάντως, ε, γενικώ θεωρώ πολύ σημαντική τη δυνατότητα που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Και επίσης συμμετέχετε στην πρώτη αυτή ευκαιρία που έχουμε για να εξετάσουμε δημοσίως τις κατεξουδότηση πράξεις και βάλαμε το θέμα αυτό στο μηνιαίο πρόγραμμα της Επιτροπής ΕΚΟΝ γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στον ρόλο και τον έλεγχο των σημαντικών αυτών νομοθετικών πράξεων. Τώρα έχουμε φυσικά ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, αλλά ως Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αν οι συντονιστές το κρίνουν απαραίτητο, τη συζήτηση για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτά λοιπόν. Η διαδικασία προβλέπει να ακούσουμε πρώτα την ομιλία του Επιτροπού Μπαρνιέ, που θα διαρκέσει γύρω στα 10 λεπτά. Κατόπιν ε, θα έχουμε 5 λεπτά ερωτήσεων και απαντήσεων. Κύριε Μπαρνιέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Καταρχήν είναι ιδιαίτερες αυτές τις στιγμές γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η τελευταία μου ευκαιρία να σας συναντήσω σε αυτήν την ολομέλεια της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα λόγια σας και για τα χειροκροτήμα για τα χειροκροτήματά σας που φυσικά επιβραβεύουν όχι μόνο εμένα προσωπικά αλλά όλη μου, όλο μου το επιτελείο, τη Γενική Διεύθυνση που συνέβαλε τα μάλα στην υλοποίηση αυτού του έργου και επίσης ε, θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο, την ποιότητα και την αγαστή συνεργασία που είχαμε με τους, ε, τα μέλη της Επιτροπής σας, ε, με τους βοηθούς, με τις διαδοχικές προεδρίες με τους συγητές, δεν μπορώ να τους κατονομάσω όλους, τους συσκιώδεις συγητές, τους συντονιστές και μια και μου δίνεται ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους βοηθούς σας που επιτελούν το έργο τους με διακριτικότητα αλλά με τεράστια ικανότητα και τους υπαλλήλους της Επιτροπής σας. Ιδιαίτερα το επιτελείο της Επιτροπής, τη Γραμματεία και τον κύριο Αντόλφο Μπαρμπέρα Δελροσάλ. Τους ευχαριστώ θερμά για την ειλικρινή και θερμή συνεργασία που είχαμε. Στις 13 Ιανουαρίου του 2010 συναντηθήκαμε για, για πρώτη φορά και στην καρδιά της κρίσης ε, και μετά το, τη συνεδρίαση του G20 με απειλές για διάλυση του ευρώ είχα χαράξει ένα χάρτη πορείας και ένα στόχο προέβλεπε ότι καμία αγορά, κανένας φορέας και κανένα προϊόν δεν μπορεί να διαφεύγει από μια δημόσια και έξυπνη ρύθμιση και από μια δημόσια εποπτεία και αποτελεσματικό έλεγχο. Χωρίς κομβασμό και διάθεση να καυχηθώ, θα ήθελα να πω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στο στόχο αυτό που δεν τον έχουμε υλοποιήσει όμως πλήρως. Πάντως η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα που ήταν η αιτία της κρίσης ε, είναι πολύ πιο ευρεία, πια πιο στιβαρή και πιο αποτελεσματική από ποτέ. Η κρίση βέβαια δεν έχει περάσει ακόμη παρόλο που η χειρότερη της φάση έχει περάσει και η οικονομική και η χρηματοπιστωτική αλλά βλέπουμε ακόμη τις ε, οικονομικές της συνέπειες ε, που πλήττουν και ταλανίζουν πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση στο, σε όλους για να κινητοποιηθούμε και θα ήθελα να σας ε, επισημάνω τρεις προκλήσεις που θα έχετε κι εσείς ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Νέα Επιτροπή. Η πρώτη πρόκληση είναι να μεριμνήσουμε ώστε να εφαρμοστούν ε, τα νομοθετικά κείμενα που έχουν ήδη εγκριθεί. Ακούγεται τριμμένο, αλλά δεν είναι. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ε, εγκρίνει 175 μέτρα επίπεδου 2, χωρίς να συνυπολογίσω τα 120 μέτρα χωρίς ε, συγκεκριμένη προθεσμία που έχουν ετοιμάσει οι Ευρωπαϊκές Αρχές Εποπτείας. Δεν πρόκειται για ε, αδύναμα μέτρα, αλλά συγκεκριμένες και ουσιαστικές προσπάθειες και μέτρα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει λοιπόν να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και εγρήγορση και χαίρομαι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εμπλακεί σε έναν λεπτομεριακό έλεγχο αυτών των κατεξουδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων, όπω είπε πριν ο προεδρό σα. Επίση. είμαι βέβαιο ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζοντας τη διαδικασία ε, εγκρίσεων του μέτρου επίπεδου 2 με διαφάνεια και με τη συνεργασία των εμπειρογνωμόνων ε, και με ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο στόχος αυτός ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα πρέπει να τηρεί κάποιε σωστέ πρακτικέ και όλα τα έγγραφα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν σταλεί στο Κοινοβούλιο. Εκπρόσωπο τη Γραμματεία Επιτροπή ήταν παρόν σε όλε τι τεχνικέ συνεδριάσει με τα κράτη-μέλη και κατά την πρώτη μηνιαία εξέταση των καταξιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων που έλαβε χώρα το Ιούλιο, οι υπηρεσίε της Γενικής διεύθυνση Εσωτερικής αγορά ε, ήρθαν για να ενημερώσουν την Επιτροπή σας ε, για την πορεία των εργασιών. Και μάλιστα οι υπηρεσίε μου είναι στη διάθεσή σας ε, και μάλιστα αύριο θα έχετε τον Γενικό Διευθυντή κύριε Γκερσόν που είναι στη διάθεσή σας. Θα έρθει και σήμερα λίγο αργότερα και προσβλέπω στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας για να ολοκληρώσουμε το ενιαίο εγχειρίδιο και μάλιστα εμπρόθεσμα. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν και Οκτώβριος ε, θα έχουν αποφασιστική σημασία γιατί τότε προβλέπεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των καταξουσιοδότηση πράξεων για τρεις εμβληματικές πρωτοβουλίες ε, της ε, επόμενης νομοθετικής περίοδου. Καταρχήν, η τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις, CRD4, προβλέπεται τον Οκτώβριο να εγκριθούν οι διεξοδικοί κανόνες για το, για το λόγο της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. Επίσης θα προσαρμόσουμε τους κανόνες της Βασιλείας για να λάβουμε υπόψη καλύτερα τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες και να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Για παράδειγμα, στην κατεξοδότηση πράξη θα μιλήσουμε για την τιτλοποίηση ε, υψηλής ποιότητας, προτείνοντας ευνοϊκή μεταχείριση των ενυπόθηκων δανείων και των ε, δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και των καταναλωτικών δανείων σε πλήρη συνοχή με την πολιτική αγορά τέτοιων ε, τιτλοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Μάριο Ντράκη φαντάζομαι θα σας ενημέρωσε προηγουμένως. Δεύτερο κείμενο αφορά τη ε, Solvency 2, Φερικαιότητα 2. Τον Οκτώβριο θα υποβάλουμε μια κατεξοδότηση πράξη που θα λάβει υπόψη τις αιτήσει, ε, τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβλέπει προσαρμογή των κανόνων ε, στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάποια μέτρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Και εδώ επίσης έχουμε την τυλοποίηση υψηλή ποιότητας με αντίστοιχο ορισμό με αυτόν που υιοθετήσαμε για το λόγο της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, LCR. Επίσης θα εγκρίνουμε ως ονόπο τις πράξεις για τον υπολογισμό των ε, εισφορών ε, των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης. Θέλουμε να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ της υποχρέωσης που έχουν όλες οι τράπεζες να συνεισφέρουν στα ταμεία εξυγίανσης όπως λέγαμε ανέκαθεν, και της ανάγκης να μειώσουμε το γραφειοκρατικό και χρηματοπιστωτικό άχθος, ιδιαίτερα για τα μικρότερα ιδρύματα. Και αυτό θα γίνει με ένα σύστημα καταποκοπήν εισφορών για, τις, για τα μικρά ιδρύματα και θα έχουμε έξι κατηγορίες μικρών τραπεζών, μικρών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα καταβάλουν καταποκοπή ποσά εισφορών που θα ανταποκρίνονται στο μέγεθός τους. Η πρότασή μας έχει στόχο να αποφύγει την διπλή καταβολή της φοράς από την ίδια τράπεζα. Δηλαδή να καταβάλει μία φορά την εισφορά ε, στο Ταμείο Εξυγίαση τη ε, Μητρική και δεύτερη φορά στην εισφορά στη χώρα της θηγατρική. Αυτό θα αποφεύγεται. Επίση ε, θα προσαρμόσουμε τις εισφορές στον κίνδυνο. Έχουμε ένα φάσμα κινδύνου 0,8 με 1,5 που είναι αρκετά περιορισμένο φάσμα Αντίθετα, τα κράτη-μέλη θεωρούν ε, ότι θα πρέπει να είναι ακόμη πιο στενό, στενή αυτή η ψαλίδα. Φαντάζομαι αύριο ήδη θα έχουμε μια συμβαστική λύση για τα θέματα αυτά και τα νομικά κείμενα θα τα οριστικοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα είμαι ακόμη στη θέση μου και θα φροντίσω να ληφθούν υπόψη και τα σχόλιά σας και τα σχόλια των εμπειρογνωμών των κρατών μελών. Επίσης ε, προσβλέπω στη συνεργασία μας ε, για να εγκριθεί η κατεξοδότηση πράξη και να δημοσιευθεί και να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2015, τότε που θα τεθεί σε εφαρμογή και η οδηγία για την εξυγίαση. Θέλουμε να υποβληθούν ταυτόχρονα οι δύο κατεξοδότηση πράξεις και για νομικούς λόγους η, εκτελεστικές πράξη, η εκτελεστική πράξη μπορεί να εγκριθεί επίσημα μόνο σε αρχές ε, του Νοεμβρίου, ενώ επί της ουσίας θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε και να δρομολογούμε από κοινού και τις δύο πράξεις. Πέραν όμως το, της εφαρμογής των ήδη ε, εγκεκριμένων κειμένων, έχουμε και ένα μια δεύτερη πρόκληση που αφορά τη συνέχιση του έργου μας ε, χωρίς ε, να χάνουμε χρόνο και να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ξεκινήσαμε. Για παράδειγμα, η ρύθμιση των δικτών αναφοράς. Γιατί είχαμε κάποιες ε, συγκλονιστικές και σκανδαλώδεις περιπτώσεις ε, χειραγώγησης ε, των, και συγκεκριμένες επιπτώσεις στα επιτόκια που έπληξαν χιλιάδες δανειολήπτες. Επίσης έχουμε την διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών ώστε να αποφύγουμε την περίπτωση τραπεζών που θα είναι υπερβολικά μεγάλες για να καταρρεύσουν ή πολύ περίπλοκες για να εξηγιανθούν ή πολύ ακριβές ε, ή δαπανηρές για να τις καθαρίσουμε ή να τις διασώσουμε με δημόσια κονδύλια. Έχουμε μάλιστα 30 τέτοιες μεγάλες τράπεζες για τις οποίες υπέβαλα πρόταση δίνοντας συνέχεια στην έκθεση Λικάνεν. Θα ήθελα να δηλώσω δημόσια ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα είναι ο κραγωνιαίος λίθος της ε, νομοθεσίας ε, για τις τράπεζες που ξεκίνησε το 2010 και νομίζω ότι είναι και η ώρα να επομιστούμε όλοι τις ευθύνες μας. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα από πλευρά μου. Επίσης έχουμε τη ρύθμιση για το, σκι... για, τις... για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, το παρατραπεζικό σύστημα, το shadow banking. Γιατί αν αφήσουμε τα παράλληλα με τις τράπεζες που υπόκειται, που στη σοβαρή ρύθμιση να έχουμε και ένα παρατραπεζικό σύστημα που θα εκφεύγει τις ρύθμισεις, ε, τι θα καταφέρουμε, απλώς να μεταφέρουμε τον κίνδυνο πέρα από τα ραντάρ της εποπτικής αρχής. Επίσης, θα πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα του shadow banking, λαμβάνοντα υπόψη τις εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης που δίνει στην πραγματική οικονομία. Αναζητούμε μια λεπτή ισορροπία που βρήκαμε κατά τη γνώμη μου στην πρόταση για τα νομισματικά ταμεία. Κάτι που είναι σημαντικό και θέλουμε να διασφαλίσουμε τον σημαντικό ρόλο της βαραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε ιδρύματα, επιχειρήσεις, ε, κρατικούς φορείς και ούτω καθεξής. Επίσης, μια άλλη σημαντική μεταρρυθμίση για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και της ανάπτυξης είναι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μακροπρόθεσμης Επένδυσης που θα γίνουν σημεία αναφοράς ε, για, κάποιες, για κάποια στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν ιδιαίτερη ρευστότητα, όπως είναι οι συμμετοχές σε μη εγγεγραμμένες εταιρείε στο χρηματιστήριο, κάποια σχέδια υποδομής και κάποια στεγαστικά ε, κατασκευαστικά προγράμματα. Θέλουμε να επενδύσουμε σε σχέδια που πραγματικά στηρίζουν την πραγματική οικονομία και θα πρέπει να βρεθούν κεφάλαια γι' αυτό. Επίσης έχουμε ένα πακέτο πληρωμών ώστε να εξασφαλίσουμε προστασία των πληρωμών μέσω διαδικτύου και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά άροντας τα εμπόδια και τους φραγμούς μεταξύ των ε, διαφόρων εθνικών αγορών εξαιτία των διαφορών που υπάρχουν στις διατραπεζικές προμήθειες. Κάτι άλλο, ένα μια τρίτη πρόκληση που είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε εύκολα. Γιατί στις χρηματοπιστωτικές αγορές υπάρχουν μερικοί ε, επιτίδιοι που αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από τους πολιτικούς. Η τρίτη μας λοιπόν πρόκληση είναι να μείνουμε σε εγρήγορση και να επαγρυπνούμε. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμής είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί λαμβάνει υπόψη την αλλαγή της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς των Ευρωπαίων. Γιατί όλο και περισσότεροι συμπολίτε μας χρησιμοποιούν τα κινητά τους ή το διαδίκτυο για να κάνουν τις αγορές τους. Και δεν καταλαβαίνουν γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στην εσωτερική αγορά. Έχουμε υπολογίσει 130 δισεκατομμύρια το χρόνο το κόστος του κατακαιρματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς των πληρωμών. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ικανότητα ε, προσερμογής μας και στον τομέα των πληρωμών. Γιατί δεν αποκλείεται στις προσπάθειές μας να ανακαλύψουμε και κάποια κενά και αδυναμίες σε ορισμένα κείμενα. Θα πρέπει λοιπόν να αναβαθμίσουμε και την, το επίπεδο φιλοδοξίας των πολιτικών συμφωνιών μας. Βέβαια η εμπειρία θα μας δείξει αν τα μέτρα που έχουμε λάβει για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά κάποιων τομέων όπως είναι στον έλεγχο όπου η περίοδος εναλλαγής των 6 ετών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατάθηκε σε 10 χρόνια, αν έχουν αποφέρει καρπούς ή θα πρέπει να συμπληρωθούν με νέα μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για την πρώτη οδηγία που εγκρίναμε την οδηγία AEFM. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τις ε, εταιρείες ε, αξιολόγησης πιστοληπτικής δυνατότητας θα πρέπει να κρίνουμε και να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο των νέων, των νέων εξουσιών της ΕΣΜΑ. Επίσης να δούμε τι γίνεται με το, τη ρύθμιση για τα hedge funds που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα στο ισχύον πλαίσιο της αυθονίας των ρευστών. Και εκεί που θα εντοπίσουμε κάποιες αδυναμίες και κάποια κενά θα πρέπει να τα καλύψουμε. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει πολυάριθμες μεταβατικές περιόδους και ρήτρες αναθεώρησης και θα πρέπει να τις να τις ενεργοποιήσουμε όπου παραστεί ανάγκη. Τέλος θα έχουμε και νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η νέα Επιτροπή και φυσικά με τις προτάσεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την όθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μερικές από τις πρωτοβουλίες αυτές έχουν προτεραιότητα, όπως η πρόληψη ε, της αντιμετώπισης των κρίσεων, ιδιαίτερα στα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή μάλλον στα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι τράπεζες. Εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση επί της ουσίας και μάλιστα σχετικά γρήγορα για να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο να αναθέσουμε σε μια ευρωπαϊκή αρχή την εξουσία επιβολή κυρώσεων με τη μορφή προστήμων οποιαδήποτε, οποιαδήποτε παραβίαση κανόνων που εξασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει από κοινού να προβληματιστούμε για τη θέση που έχει η Ευρώπη στις, στους διάφορους λογιστικούς κανόνες σε όλες ε, τις ε, συνεδριάσεις που έγιναν τελευταία πέντε χρόνια ε, θέσαμε το θέμα αυτό αλλά δεν βρήκαμε μια σωστή ισορροπία σε διεθνές επίπεδο για την κατάρτιση τέτοιων κανόνων. Δεν έχουμε πετύχει την επιθυμητή σύγκληση, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί δεν ξέρω αν ποτέ οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεχτούν ποτέ αυτή τη σύγκληση των κανόνων στα θέματα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, νομίζω ότι υλοποιήσαμε μια στιβαρή μεταρρύθμιση άνευ προηγουμένου, ήταν σχεδόν επαναστατική για πολλές τράπεζες και δείξαμε το καλό παράδειγμα και στον κόσμο. Οπότε είναι θέμα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που λάβαμε από κοινού στο G20 και στη σχέση μας με τις τρίτες χώρες είμαστε έτοιμοι, χωρίς όμως να είμαστε και αφελείς ταυτόχρονα, να συνεργαστούμε με τις τρίτες αυτές χώρες, υπό τον όρο όμως ότι και οι τρίτες χώρες, ιδιαίτερα οι Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά όχι μόνο, θα υιοθετήσουν κανόνες αντίστοιχους ε, ή εφάμιλους με τους δικούς μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να πληρούνται τέσσερις προϋποθέσεις. Πρώτον, εμείς από πρώτοι από όλους να εφαρμόσουμε με σοβαρότητα τις μεταρρυθμίσεις μας. Δεύτερον, να εδραιώσουμε τη διεθνή συνεργασία στα πλαίσια του G20 και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τρίτον, να είμαστε ενωμένοι και στιβαροί, να δείξουμε πυγμή στις διμερείς συζητήσεις μας χρησιμοποιώντας όλους τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας συμπεριλαμβανομένης και της ε, ε, χορήγησης ή ε, μη χορήγησης της αμοιβαιότητας και το TTIP, τις Διατλαντικές Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης για, τις, για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε διαφάνεια στις σχέσεις με, τους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι οι κύριοι εταίροι μας. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει τα όρια. Λοιπόν, εφαρμογή των λιμένων αποφάσεων, συγκεκριμενοποίηση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, εγρήγορση, δυνατότητα προσαρμογής, προσαρμοστικότητα είναι σημαντικές προκλήσεις που το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τις αναλάβουν από κοινού με το Συμβούλιο. Πάντως αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και είμαι υπερήφανος για τη συνεργασία που είχαμε και σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, για την παρέμβαση αυτή και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για τη συζήτηση με πρώτο τον Μάρκους Βέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο πρόσωπό σας για τη δουλειά που κάνατε, που ήταν ε, στο έργο τεσσάρων επιτρόπων με τη νέα κατανομή χαρτοφυλακίων στην Επιτροπή. Προφανώς σας παρακαλουθούμε με μεγάλη προσοχή και προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην προσεχή θητεία πολλά θέματα νομοθεσίας από το επίπεδο 1, level 1, στο επόμενο επίπεδο και φαντάζομαι ότι θα πρέπει και εσείς να λύσετε κάποια ζητήματα μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Δεν μπορείτε δηλαδή να επαναπευθείτε στις δάφνες σας μέχρι την 1η Νοεμβρίου που θα αναλάβει η νέα επιτροπή θα έχετε ζητήματα να επιλύσετε και κυρίως ε, την πρόοδο της Τραπεζικής Ένωσης του μηχανισμού, ε, χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ε, μηχανισμό χρηματοπιστωτικής εποπτείας, όλα αυτά που αποτελούν αξιολόγηση του κινδύνου και όπου δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, για να το πω επίοικος, από τις εξελίξεις. Δεν πρέπει δηλαδή να αγνοούμε παράγοντες οι οποίοι μπορεί να ενισχύουν τον κίνδυνο με τη νέα νομοθεσία. Τις λεπτομέρειες της γνωρίζετε, έχει προηγηθεί η ανταλλαγή επιστολών, συζητήσεις, έχουμε ζητήσει πολλές φορές μέσα στο μήνα ή έστω προς αρχές του Οκτωβρίου να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έχουμε την ευκαιρία ελπίζουμε να συζητήσουμε για να αποστείλουμε και εμείς από πλευράς μας ένα σαφές μήνυμα. Και όπου υπάρχουν κίνδυνοι πρέπει αυτοί κατά τον υπολογισμό της συμβολής, της συμμετοχής να ε, υπολογίζονται με πολύ μεγάλο προσεκτικό. Ξέρετε ότι το netting των παραγόγων για μας δεν είναι ικανοποιητική λύση, δεν περιορίζει τον κίνδυνο και ιδιαίτερα για τα συστήματα τα οποία ε, μπορεί να αποτελούν συσχετισμούς ευθύνης και αυτορυθμίζονται ή αυτοαποκαθιστούν την ασφάλεια για μας δεν είναι η λύση. Πάντοτε θέλουμε μια προσέγγιση που να στρέφεται και προς τα προβλήματα των μικρότερων τραπεζών. Πρέπει λοιπόν σε επόμενες ημέρες ή εβδομάδες αναλόγως δυνατότητές σας να δούμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις από τις υπηρεσίες σας. Ευχαριστώ. Κύριε Βαρνιέ. Όπως θέλετε εσείς, θέλετε, έχετε πέντε λεπτά για την κάθε ερώτηση, επομένως ο κύριος Βαρνιέ. Ναι, βεβαίως και είμαι έτοιμος να απαντήσω στην ερώτηση ειδικά για τον παράγοντα κίνδυνο. Φαντάζομαι ότι και άλλοι βουλευτές μπορεί να έχουν το ίδιο θέμα. Για να διευκολύνω λοιπόν τη συζήτηση, προτιμώ να ακούσω και άλλες ερωτήσεις. Εάν συμφωνεί και ο Μάρκο. Καλώς τότε θα δώσω το λόγο στην Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ και πάλι. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ για την καταπληκτική δουλειά που έχετε καταφέρει να κάνετε με όλους σας, με σας το επιτελείο. Μια ομάδα πάντα διαθέσιμη, πολύ αποτελεσματική και που πιστεύω σε μια δύσκολη για τη συλλογική μας ζωή και τη ζώνη του ευρώ περίοδο μας επέτρεψε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστώ πολύ που στην τελευταία αυτή συνεδρίασή μας ε, φέρατε προς συζήτηση θέματα που μπορούν να αποτελέσουν κατά την άποψή σας συμβουλές για το Κοινοβούλιο και για τον διάδοχό σας. Θέματα που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε κατά την πρόοδο στις εργασίες μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις, στις οποίες θέλω τη γνώμη σας και τις προτάσεις σας. Πρώτη, στο θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα πρόοδου απρόβλεπτο ακόμη πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Δεν υπήρχε καν η δυνατότητα να φανταστεί κανείς, να διανοηθεί κανείς ότι θα φτάναμε σε μια τραπεζική ένωση. Τώρα πια έχει γίνει το πιο περίπλοκο βήμα, ωστόσο από το σενάριο αυτό βλέπουμε να έχει χαθεί ένα στοιχείο, κοινή εγγύηση καταθέσεων. Θέλω το σχολείο σας λοιπόν, γιατί υπήρχε μια κοινή πολιτική δέσμευση το 2012 με τα τρία στοιχεία, την εποπτεία, την ε, εκαθάριση, την εξυγίανση και την κοινή εγγύηση των καταθέσεων. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά προχωρούν σε σταδιακές φάσεις και σε ε, αλλεπάλληλες φάσεις, αλλά έχει χαθεί η κοινή εγγύηση καταθέσεων. Άλλωστε το και εσείς την αναφέρατε. Τι έγινε λοιπόν, εξαφανίστηκε για τον κοινό μηχανισμό καθάρισης αυτό, αυτή η δουλειά συνεχίζεται με τις υπηρεσίες σας ε, για τις καταξουσιοδότητες συμπράξεις, το είπατε και εσείς. Ωστόσο θέλω τη γνώμη σας ως προς την διακυβερνητική συμφωνία. Αν βλέπετε κάποια κινητικότητα, αν έχει προσδιοριστεί χρονοδιάγραμμα για την ε, επικύρωση της διακυβερνητικής συμφωνίας με βάση την οποία θα, διατεθούν οι συνεισφορές, η μεταφορά δηλαδή από τις τράπεζες προς, από τον κορβανά τον κρατικό προς το κεντρικό ταμείο για να το πω έτσι. Και επίσης πολύ φοβούμαι ότι λησμονήθηκε στην πορεία αυτή μια υπόσχεση που είχε δοθεί κατά τρόπο τυπικό μια δέσμευση σοβαρή από πλευράς του Συμβουλίου, ότι δηλαδή θα αναζητούσε μια πιστοτική γραμμή για το Ταμείο Εκαθάρισης για την αρχική του φάση, ώστε να του δώσει μια κάποια βαρύτητα περισσότερη μόχλευση για να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί και να φέρει αποτελέσματα στην πρώτη οκταετία. Και έτσι βέβαια έχουμε και το επόμενο θέμα που έθιξε και ο Σάνελφος Φέρμπερ και που όλοι μας συζητούμε. Κεντρικό ζήτημα λοιπόν εδώ είναι εάν τα ζητήματα που είχε επισημάνει σε πρώτο επίπεδο, στην ε, πρώτο επίπεδο νομοθεσία το Κοινοβούλιο, έχουν πράγματι ληφθεί υπόψη και αντικατοπτρίζονται στις λεπτομέρειες και αν ο παράγων κινδύνου είναι όντως ο πιο ουσιαστικός. Δεν θα υψαλθώ σε λεπτομέρειες, τα γνωρίζουμε όλοι. Αν θέλετε λοιπόν να μα δώσετε κάποια πιο ε, επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και έτσι θα μπορέσουμε, αν το πράξετε, να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις προσεχείς συνεδριάσεις με τον διαδοχό σας, με τους διαδόχους Ευχαριστώ πολύ Λίζα. Συντηρητικοί μεταρρυθμιστές, Johann van Φαν-Οβερτφέλτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παρνιά που είστε εδώ και για τη σπουδαία σας δουλειά για την Τραπεζική Ένωση. Έχω δύο ερωτήσεις και οι δύο σχετίζονται με τις συμβολές ε, που θα κάνουν οι τράπεζες. Η πρώτη είναι η εξής. Πώς θα εξασφαλίσει η Κομισιόν ότι δύο ε, τράπεζες που θεωρούνται μικρές ε, από, με βάση τον ορισμό της ΕΜΠΕΡΔ και που έχουν ε, τον ίδιο προφίλ κινδύνου δεν θα καταλήξουν να πληρώνουν διαφορετικές συμβολές απλά και μόνο επειδή μια από αυτές έχει έδρα σε μια χώρα που είναι στη διαδικασία υπερβολικού χρέους, ενώ οι άλλοι όχι. Δηλαδή το μοντέλο υπολογισμού υπολογίζει τον κίνδυνο της οικονομίας εντός της οποίας λειτουργεί η κάθε τράπεζα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση, πώς θα εξασφαλίσετε ε, ισότιμο πεδίο για τις συμβολές που θα καταβάλουν οι τράπεζες ίδιου μεγέθους και ίδιου προφίλ κινδύνου στην Ευρωζώνη και εκτός της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Thank Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλντε, Νίλ Τόρβαλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ Επίτροπε Μπαρνέ που είστε σήμερα εδώ. Στην αναρτήριά σας εισήγηση μιλήσατε για ένα εγχειρίδιο, ενιαίο εγχειρίδιο Ε, Ποιε είναι οι δυνατότητες για κατακαιρματισμό και πώς θα αποφευχθούν. Σήμερα ορισμένα κράτη δίνουν φοροαπαλλαγές για τι ε, τις τραπεζικές ε, Συνήθω Συνήθως μιλάμε για την ανάγκη να μην μετακυλίονται τα προβλήματα των τραπεζών στους φορολογούμενους, όμως μετά από την πίσω πόρτα κάποιες χώρες εξακολουθούν να το πράττουν αυτό. Γαλλία, Βέλγιο και Σουηδία το κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μετακυλείται το κόστος ε, στους φορολογούμενους, γιατί αυτό στρεβλώνει και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις τράπεζες. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν έχετε κάποιο σχέδιο για να το αντιμετωπίσετε αυτό, η Κομισιόν ή όχι. Έχετε κάποιο σχέδιο δηλαδή για εναρμόνιση σε αυτό το τομέα ώστε να επικρατούν οι ίδιοι όροι για όλους. Γιατί πολύ συχνά εμείς οι πολιτικοί μιλάμε για ίσους όρους για όλους ακόμα και αν στη συνέχεια μετά ορισμένοι προσπαθούν πάλι να παρακάμψουν τους κανόνες. Σας ευχαριστώ για την ΚΟΥΕ, ο κύριος Φάμπιο Ντεμάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαρνιέ. Και εγώ θα ήθελα από πλευράς μου να σας ευχηθώ κάθε καλό για την ε, περίοδο μετά την αποχώρησή σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην αρχή της παρέμβασης είπατε ότι ε, έχει γίνει πιο αποτελεσματική η ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών. Επιτρέψτε μου όμως να παραπέμψω σε ένα άρθρο του Μάρτιν Γούλφ από Financial Times, ο οποίος Αναφέρεται σε πράξη στο Dort Act ε, υπό τον Ομπάμα με 70 τόσες σελίδες και άλλη νομοθεσία με 30 τόσες σελίδες. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν ξέρω πόσες σελίδες μετρά, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο αποτελεσματική και είμαι πολύ επιφυλακτικός όταν βλέπω ότι έρχονται λόμπι, από την ε, ε, City of London για να αναλάβουν καθήκοντα ακριβώς στον χώρο της ε, διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεν ξέρω εάν η Τραπεζική Ένωση αποτελεί μια λύση καλή, μια λύση που να σέβεται τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και να τον προστατεύει. Δεν ξέρω εάν το Ταμείο Καθαρίσης με τα 55 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να δώσει, με τα 155 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να δώσει τις λύσεις που περιμένει ο φορολογούμενος και είναι σοβαρή απάντηση, αλλά θέλω να ρωτήσω τα εξή. Κατά τη δική σας εκτίμηση, αυτή, τα, τα too bank to fail, η ιδέα δηλαδή ότι έχουν ε, αυτόματα κάποιο πλεονέκτημα να χρηματοδότηση ορισμένε μεγάλες τράπεζες, ε, έχει περιοριστεί ή μήπως η μηπω η συγκεντρωση στο τραπεζικό τομέα έχει αυξηθεί αντίθετα. Δεύτερον, Πιστεύετε ότι στο Ταμείο Εκαθάρισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες μορφές τραπεζικές όπως τα ταμιευτήρια, τα, τα γερμανικά, η Σπάρκας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να τηρήσει τον κανόνα των ιδίων κεφαλαίων για την εγκατάσταση αλλοδαπών τραπεζών που είναι πιο αυστηρό στις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο Φίλιπ Λαμπέρτς. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι έχω την ίδια επιχειρηματολογία όπως και ο Φάβιο Ντεμάζ. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν τα όσα είπε. Κύριε Μπαρνιέ, είστε ένας ε, πολύ εξαιρετικός άνθρωπος γιατί έρχεστε από την ε, τελευταία πραγματική μοναρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά μας δείξατε μια όρεξη πολύ μεγάλη και μια αγάπη για τον κοινοβουλευτισμό που σίγουρα δεν σας έρχεται από τη Γαλλία. Ε, έχετε δώσει μεγάλη σημασία στο Κοινοβούλιο, δεν έχετε προσποιηθεί και μόνο και μόνο γι' αυτό σας ευχαριστώ. Ο Φάβιο αναφέρθηκε στον όγκο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και κατά τη γνώμη μου αυτός ο όγκος αποδίδεται στο γεγονός ότι όσο πιο περίπλοκη είναι μια νομοθεσία τόσο περισσότερο προσφέρει δυνατότητες παράκαμψης του πνεύματός της. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο με το κείμενο του πρώτου επίπεδου, αλλά και με τον όγκο, το είπατε και εσείς ο ίδιος, με τις νομοθετικές πράξεις δευτέρου επίπεδου που θα χρειαστεί να εγκρίνουμε σε αυτή τη θητεία. Η πρώτη προβληματική είναι η BERD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης για την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίαση, με συγχωρείτε. Ε, και θα πρέπει εμεί αυτό να συμβάλλουμε και να συμβάλλουν οι τράπεζε. Αυτέ που αντιπροσωπεύουν το 85% θα συμβάλλουν κατά το 98% του ε, συνόλου, δηλαδή περίπου την αναλογία του. Είτε είναι 1,6 μέχρι 3, ό,τι να είναι. Ο παράγοντα κίνδυνο παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο στη συμβολή των τραπεζών. Και γι' αυτό αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε και αυτό προέρχεται από τις μεγάλες γαλλικές τράπεζες και τις μεγάλες γερμανικές, ιταλικές και ισπανικές τράπεζες. Είναι οι συστημικές τράπεζες που επιθυμούν να ξεφορτωθούν τα χρεόγραφά τους. Έπειτα, ε, αναλογία Ε, ε, ε, ρευστότητες με, κεφα... με κεφάλαια, με εγγύησεις στο πλαίσιο της οδηγίας ΕΡΔΕ. Εδώ θέλει θέλουμε να προσθέσουμε τα καλυμμένα ομόλογα και τα ABS για τα οποία μιλάμε διαρκώς εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και, όμως η νομοθεσία λέει πως αυτά τα δύο στοιχεία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν ως ρευστά ενεργητικά παρά μόνο αν αναγνωρίζονται ως τέτοια από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αγορά. Όμως αυτό δεν ίσχυε και η Κομισιόν θέλει αυτό να το παρακάμψει. Γιατί λοιπόν εκ νέου θέλουμε να ελαφρύνουμε ε, ε, κανόνες που ο νομοθέτης ήθελε αυστηρά στις πράξεις δευτέρω επίπεδου, το ίδιο και για την φεργιότητα 2. Και εδώ εκ νέου αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το παράθυρο Ισχύει μια ευνοϊκή διάθεση σε σχέση με τα ABS, θέλοντα να μειώσουμε το επίπεδο το παρέτου του κεφαλαίου για να καλυφθούν οι κίνδυνοι που τα συνοδεύουν και αυτό με τον κίνδυνο να αποδιαρθρωθεί η σχετική αυστηρότητα του νομοθέτη μέσω των πράξεων του δευτέρου επίπεδου που κατά κάποιο τρόπο αποδυναμώνουν το σύνολο. Πολύ θα με λυπούσε λοιπόν εάν μετά από το δικό σας πέρασμα ή στο τέλος της θητείας σας τελικά ήδη να αρχίζουμε μετά από πίεση των μεγάλων ε, χρηματοπιστωτικών ομίλων να αποδυναμώνουμε, να αποδυναμώνουμε αυτό που ήταν εν μέρη δικό σας έργο. Από την ευθυντή δεν έχω δει κανένα αίτημα. Θέλει κάποιο συνάδελφο να πάρει το λόγο. Όχι. Οπότε τότε μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους ομιλητές, συντονιστές, εκπροσώπους των ομάδων που δέχτηκαν να γίνει ομαδοποίηση των ερωτήσεων γιατί βλέπουμε ότι επανέρχονται τα ίδια ζητήματα για τον Μάρκος Βέρπερ και τη Λίζα, Ελίζα Φερέιρα. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να τεθεί σε ισχύ η Τραπεζική Ένωση. Κύριε Φερέιρα, εσείς είπατε ότι ήταν απροσδόκητο, έτσι δεν είπατε. Αναπάντεχο. Τα θυμάστε όλοι μαζί ήμασταν στις αρχές εκείνες όπου είχα πει ότι σκοπεύω να θεσπίσω τις αρχές ε, ευρωπαϊκής εποπτείας όπως τις είχε προβλέψει η έκθεση Ντελαροζιέρ. Βεβαίως και είχαμε και ιδέες για πιο μεγάλα βήματα, πιο σημαντική πρόοδο, αλλά ήταν αδιανόητο το 2010 το να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μέσα στη ζώνη του ευρώ σε μια ομοσπονδιακού, ομοσπονδιακή στόχευση ένωση των τραπεζών ήταν αδιανόητο και όμως κατέστη δυνατό και χάρη στις προσπάθειες των ε, πολιτικών ομάδων του Προέδρου Μπαρόζου, του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας. Ε, όλοι από το 2012 και μετά κάναμε προσπάθεια και ενώσαμε και δώσαμε τελικά την ε, λύση της Τραπεζικής Ένωσης. Και βέβαια σε αυτό η εποπτεία και η επαγρύπνηση του Κοινοβουλίου είχε κέριο ρόλο. Για τα άλλα ερωτήματα, ίσως να μην μπορούσαν να απόλυτα ικανοποιητικέ απαντήσεις με τις λεπτομέρειες. Αύριο με τον κύριο Κερσάν θα έχετε με τον Γενικό Διευθυντή, δηλαδή τη δυνατότητα να δείτε τις λεπτομέρειες. Σας παρακολουθεί, βρίσκεται εδώ. Θα ε, μπει στο δυνατό βαθμό στις λεπτομέρειες. Για τον παράγοντα του κινδύνου όμως που αναφέρθηκε ο κύριος Μάρκους Βέπερ, ήδη έχουμε την έννοια του risk sensitive ε, γιατί οι ίδιοι πόροι δεν υπολογίζονται με αυτήν την έννοια. Δηλαδή όσο πιο πολλούς έχει μια τράπεζα τόσο, πιο τόσο θα υπολογίζεται μικρότερη συνεισφορά σε σχέση με τον ισολογισμό της. Άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν χειραγωγήσεις στον τομέα αυτόν. Για τον πρόσθετο όμως παράγοντα κινδύνου με βάση την οδηγία Αμπέρντε που αναφέρθηκε νωρίτερα και που έχουμε συζητήσει, έχουμε προτείνει τέσσερις πυλώνες ως βάση εργασίας. Έκθεση στον κίνδυνο με 50% στάθμιση και τέσσερις δείκτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το RWA, το risk rate, το ποσοστό ιδίων πόρων, αλλά και σε ισότιμη βάση και ως εκ τούτου με πολύ μεγαλύτερη στάθμιση από τις CRD4, την μοχλευτική ικανότητα και εν τέλει τους ε, διαθέσιμους για τον Μπέιλιν πόρους. Στο δεύτερο έχουμε την σταθερότητα ή την διακύμανση των ε, πόρων με, τα, με τις δύο αναλογίες ε, ρευστότητας του CRD4. Μετά έχουμε την προβλεψιμότητα του δημοσιονομικού του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την έκθεση σε άλλους φορείς. Μετά έχουμε τις λοιπές δραστηριότητες με στάθμιση 20%, το trading, τις κρατικές ενισχύσεις κτλ. Ε, Πυλώνας μάλιστα που είναι δύσκολο να βαθμονομηθεί, να υπολογιστεί εκ των προτέρων το μέγεθός του και έτσι αφήνουμε μεγαλύτερο περιθώριο αξιολόγησης στις αρχές εκαθάρισης. Είπατε, αλλά νομίζω και το ανέφερα και εγώ, ότι υπάρχουν τρεις θεωρίες ως προς ε, την ε, ψαλίδα του κινδύνου από το 0,8 στο 1,5. Η βασική συνεισφορά, το είπα και νωρίτερα, είναι risk sensitive. Το ανέφερα στην προηγούμενη, προηγούμενη μου απάντηση. Μια απλή φόρμουλα, ένας απλός τύπος δηλαδή που θα είναι δύσκολο να χειραγωγηθεί. Ξέρω ότι σας φαίνεται υπερβολικά στενή αυτή η ψαλίδα, αυτό το περιθώριο, αλλά σας το επαναλαμβάνω, γιατί ήταν και συμβασμός μεταξύ των δύο συνομοθετικών αρμοδίων αρχών, δηλαδή του Συμβουλίου και ημών. Για το, στο Συμβούλιο υπήρχαν κάποιοι που ήταν υπερβολικά διστακτικοί και χρειάστηκε να καταλήξουμε στο, στο συμβασμό αυτόν. Η κυρία Φερέιρα αναφέρθηκε στην εγγύηση των καταθέσεων. Όντω η νέα επιτροπή θα χρειαστεί να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Εγώ υπενθυμίζω ότι αποτελεί στοιχείο του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα το πολύ σημαντικό αυτό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης δεν πρέπει να λησμονηθεί. Έχουμε όλοι μαζί προχωρήσει σε πολλούς συμβασμούς. Δεν ήταν όλοι πάντοτε ικανοποιητικοί. Αλλά πιστεύω ότι η νέα Επιτροπή θα πρέπει πλέον να αναλάβει τις ευθύνες της. Ίσως μπορώ και γραπτός να σα απαντήσω κύριε Φερέιρα για το χρονοδιάγραμμα της επικύρωση, γιατί δεν θέλω να σα δώσω πρόχειρες ε, απαντήσει. Έχω μια αμφιβολία ως προς τις προθεσμίες και προτιμώ να μην κάνω δηλώσει δημόσιες που ενδεχομένω να με δέσμευαν. Ε, και αυτό προτιμώ να το επαληθεύσω με το Συμβούλιο πρώτα και μετά να απαντήσω. Επίση, και αυτό νομίζω έρχεται και να συμπληρώσει την ερώτηση του κυρίου Ντεμάση, Είπατε κάτι για, την, ε, ικανότητα, για το δυναμικό του Ταμείου Καθαίρεση. Είπε ο κ. Δεμά ότι τα 55 εκατομμύρια δεν είναι επαρκή. Είπε η κυρία Φεραίρα ότι θα χρειαστούν και άλλα μέσα. Βεβαίω θα πρέπει να δώσουμε τα μέσα δράση στο Ταμείο Καθάρισης ώστε να μπορεί να λαμβάνει τι αποφάσει και να τι υλοποιεί, ώστε να καταστεί αξιόπιστο από την πρώτη στιγμή λειτουργία του. Και το Ταμείο, εάν χρειαστεί, εάν παραστεί ανάγκη, θα πρέπει να είναι σε θέση και να αντλήσει από τι αγορέ κεφάλαιο προκειμένου να έχει αρκετή ε, βάση ξεκινώντας. Ο κύριος Φανόφερτ ε, φαίνεται έχει αποχωρήσει. Είχε δύο ερωτήσεις. Θα απαντήσω λοιπόν λακωνικά. Κύριο Λάμπερτ, ε, αναγνώριζε ότι γνωρίζω πολύ καλά τι δεσμεύσει έχουν οι βουλευτέ ε, πάντα ανηλυμένε υποχρεώσει Το δέχομαι. Λοιπόν, για το ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ζώνη του ευρώ ω ένα σύνολο. Μα ακριβώ αυτό ήταν ο στόχο μα με την ε, Τραπεζική Ένωση. Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε διαφορετικό παράγοντα κινδύνου για το κάθε κράτο, γιατί αυτό θα αντέβαινε ακριβώ στο χαρακτήρα και στο, στη στόχευση τη Τραπεζική Ένωση. Το γεγονό ότι εφαρμόζουμε την συνεισφορά στο επίπεδο της Τραπεζικής Ένωσης. Ήδη θα έχει επιπτώσεις προς την εθνική συμβολή και θα πρέπει στην εκτελεστική πράξη να εξισορροπηθούν οι δύο αυτές έννοιες. Το μελετάμε. Βάση Τραπεζικής Ένωσης και εθνικές αρχές. Αυτά λοιπόν είχα να πω για τον κύριο Φανόβερτσφελτ. Ο κύριος Κόβατς μου έστειλε σε κάποιες ερωτήσεις στις οποίες αποδίδω μεγάλη σημασία το ζήτημα του βασικού τραπεζικού κώδικα, το ζήτημα της διαφάνειας για τον πιο ευάλωτο φορολογούμενα, το ζήτημα της διαφοράς μεταχείρισης καταναλωτών πολιτών. Παραπέμπω λοιπόν στο κείμενο αυτό το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί και το οποίο ξέρετε ότι αντιμετώπισε πολλές πιέσεις από τα λόμπι. Χρειάστηκε λοιπόν να κρατήσω αντιστάσεις και μαζί με έναν πρώην συνάδελφο τον κύριο Κλούτε πήραμε αποφάσεις για την ε, τραπεζική κινητικότητα, για την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό για τον κάθε πολίτη, γιατί ξέρετε αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, σε ορισμένες υπάρχει, αλλά όχι πάντα. Κύριε Βάλτς υπάρχει το ζήτημα και της συγκρισιμότητας των ε, τελών το οποίο, η οποία θα καταστεί υποχρεωτική για την κάθε χώρα. Δηλαδή θα υπάρχει ένας πίνακας που θα καθιστά δυνατή την ε, σύγκριση. Η διαφάνεια νομίζω ότι είναι η βασική αρχή, η βασική προϋπόθεση της ευθύνης. Αν έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε με έναν πίνακα τα τέλη, το κόστος, ε, αν υπάρχουν ε, επιπλέον επιβαρύνσεις κόστος επιπλέον, μπορούμε να κρίνουμε τι προτιμάμε. Αυτό λοιπόν. παράλληλα και με την παρακολούθηση από τις αρμόδιες επιτροπές ε, οι οποίες θα ε, προστατεύουν τον καταναλωτή από την υπερβολική χρέωση και τα υπερβολικά τέλη. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεμάση για τις ε, ευχές του για το, για το περαιτέρω. Δεν μπαίνω σε μια επόμενη φάση του δημόσιου βίου μου χωρίς να έχω αντλήσει διδάγματα από την τελευταία πενταετία. Εγώ προσωπικώς έχω ο άνθρωπος, έχω διδαχθεί πολλά και περνώ σε μια επόμενη φάση της πολιτικής μου ζωής στη Γαλλία με τη νέα εμπειρία που έχω αποκομίσει μαζί σας και πολλές φορές χάρη σε σας. Και θέλω να με πιστέψετε όταν λέω ότι το κλειδί είναι τα χρηματοοικονομικά να την χάνουν διαχειρίσεως ορθολογικής και διαφανούς προς το συμφέρον της πραγματικής οικονομίας πάντα και όχι αυτό που έχει γίνει μερικές φορές μέχρι τώρα εις, ε, όφελο ε, του, του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά εις βάρος της πραγματικής οικονομίας. Τον διάδοχό μου δεν θα τον κρίνω προφανώς. Καλό όμως εσάς να τον κρίνετε και βάσει βέβαια αρχικά των δηλώσεών του αλλά και ε, στη συνέχεια βάσει των πράξεων του και όχι βάσει της εθνικότητάς του. Ξέρετε ότι και εγώ πολλές φορές έπεσα θύμα δικών προθέσεων από διάφορες εφημερίδες κυρίως, ε, γιατί ήμουν Γάλλο. Για κοιτάξτε στα αρχεία των εφημερίδων. Με είχαν χαρακτηρίσει ορισμένοι ως τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στην Ευρώπη. Εγώ είπα κρίνεται με από τις πράξεις μου. Ε, τίποτα άλλο δεν μπορώ να ευχηθώ στους, ε, σε όποιον πάρει τώρα την σκητάλη. Για τα 55 δις σας απάντησα. Για την συμφωνία TTIP έχω εκφράσει την επιθυμία αλλά παραμένουν πολύ ε, αρνητικοί οι Αμερικανοί. Το ζήτημα, η διαδικασία πάνω απ' όλα, όχι η ουσία, η διαδικασία ε, να προχωρήσει μέσα από μια συμφωνία και μια μέθοδο κοινή μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων, όχι για να πέσουν οι προδιαγραφές ε, και το επίπεδο των απαιτήσεων το, των αντίων. Το έχω επαναλάβει αυτό πολλές φορές και σε επίπεδο και, και απευθυνόμενους Αμερικανούς εταίρους. Αλλά για να δώσουμε νέα δυναμική σε όλα τα φόρουμ, σε όλα τα κέντρα συζητήσεων που επιμέρους αναπτύσσονται σε τομεακό επίπεδο και τα οποία πολλές φορές δεν λειτουργούν αρκετά αποτελεσματικά στις ΗΠΑ. Εγώ έχω, συμμετάσχει, έχω, έχω παρακολουθήσει διαφορετικά φόρουμ, παραδείγματι για τη χρηματοοικονομική ε, ρύθμιση, διακυβέρνηση. Θα ήθελα να ενισχυθεί περισσότερο αυτός ο τομέας της και να υπάρξει μια διαλειτουργικότητα πλήρης, ε, σαφής, αποτελεσματική, δηλαδή να ε, αλληλεπιδρούν οι δύο, τα δύο εγχειρίδια, τα δύο σύνολα κανόνων από τη μία και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Κύριε Ντεμάση, η οικονομική διαχείριση είναι πιο αποτελεσματική. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να επαναπάβομαι σε δάπνες, δεν έχει τελειώσει η δουλειά, εσύ, η δική σας δουλειά δεν έχει τελειώσει φέτος ή του χρόνου, θα πρέπει να προχωρήσετε. Εμάς μας πήρε μέχρι και τέσσερα χρόνια η πρόοδος στα νομοθετήματα αυτά, χρειαζόμαστε πιο απαιτητικούς κανόνες, χρειαζόμαστε αρχές εποπτικές, χρειαζόμαστε ιδίους πόρους που έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Αυτά όλα έχουν προχωρήσει. Έχουν όμως αποτραπεί όλοι κίνδυνοι. Η απάντηση είναι όχι. Εξού και καλώ σε επαγρύπνηση και λέω εγώ ότι θα πρέπει να προσαρμόζεται το νομοθετήματο που διαπιστώνονται ε, ελλείμματα ή παραθυράκια μέσα από τα οποία θα μπορούσε να διαφύγει κανεί. Για το ζήτημα των πολύ μεγάλων τραπεζών περίμενα ότι θα ακουστεί μια τέτοια ερώτηση, έστω και αν κάποιοι είχαν διατυπώσει την εποχή εκείνη επικρίσεις σημαντικές, τις οποίες βεβαίως έτεινα ευήκονους, αλλά εν τέλει, και το ερώτημά σα είναι εάν αρκεί αυτό, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να θέσει κανεί στην αρχή τη διαδικασία. ούτε καν στα μισά της διαδικασίας της ρύθμισης. Μαζί με τον κύριο Λίκανεν, ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το θέσαμε το ερώτημα, διαρωτηθήκαμε αν αρκεί, αλλά περισσότερο το 2013 όταν είχαμε μια σαφέστερη εικόνα για όλα τα νομοθετήματα που θα φορούσαν τις τράπεζες, ε, με τις εγγύησεις καταθέσεων, με την εκαθάριση, την εποπτεία, ε, την ε, διακυβέρνηση, όλα αυτά τα ζητήματα τα θέσαμε. Και η απάντηση δική μου ήταν εφόσον εφαρμοστούν τα νομοθετήματα, βεβαίως και αρκεί για τις περισσότερες τράπεζες, εάν όχι αρκεί μόνο για λίγες. Για τις πολύ μεγάλες, too big to fail, too costly to resolve και όλα αυτά, υπό αυτές που είναι πολύ κοντά στον κρατικό μηχανισμό κτλ. Νομίζω ότι τα ερωτήματα πρέπει να τα θέσουμε στην φάση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των τραπεζών που υποβάλαμε. Αυτά. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τον Φίλιπ Λαμπέρτς και τις θέσεις του για την, ε, για την μοναρχία στη Γαλλία. Κοιτάξτε, εγώ είμαι του κοινοβουλευτικού συστήματος ανέκαθεν. Ήμουν βουλευτής στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, είχα την τιμή να εκλεγώ και ευρωβουλευτής αρκετό καιρό μέχρι που ανέλαβα κάθε... πρωτού μάλλον αναλάβω καθήκοντα. Επιτρόπου έχω κάθε σεβασμό στον κοινοβουλευτισμό κύριος Λομπέρτς αλλά και όλοι όσοι εκ των συντονιστών τοποθετήθηκαν πριν από εσά νομίζω ε, ότι μπορώ να περιμένω αυτό το σεβασμό και την ε, προσδοκία από το σεβασμό από το Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε στην αναλογικότητα νωρίτερα και τις συνέπειες για τις μικρότερες τράπεζες ε, που προκύπτουν από την εισφορά. Προσπαθώ να βρω την χρυσή τομή, μια ισορροπία λεπτή. Το είδαμε, σας το εξήγησα και με όλα τα νομοθετήματα. Ε, προσπαθώ λοιπόν με το σύστημα της καταποκοπήν συνεισφοράς για τις μικρές τράπεζες, οι οποίες θα καταβάλουν ένα ποσό καταποκοπήν ανάλογα του μεγέθους τους και με βάση τις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις μας, υπενθυμίζω το μεταξύ ότι η πρόταση αυτή, η μέθοδος που προτείνουμε, οδηγεί σε συγκεκριμένα ποσά, που θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, οι τράπεζες οι οποίες έχουν το 85% του ενεργητικού της ζώνης ευρώ θα έχουν συνεισφορά κατά 80% τουλάχιστον του συνόλου των συνεισφορών. 90%. Και όταν έχουν πάνω και 50% των τραπεζικών ιδρυμάτων θα έχουν το ειδικό καθεστώς που αφορά τα μικρά τραπεζο... τραπεζικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, αυτά λοιπόν θα έχουν μία μείωση της τάξης του 70% των ε, συνεισφορών τους στη ζώνη του ευρώ. Βρήκαμε και νομίζω πλησιάσαμε αρκετά ε, στην ε, αναζήτηση αυτή ενός επίπεδου αναλογικού στη συνεισφορά ανάλογα και με τον κίνδυνο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Έχω πέντε ακόμα μιλήτες Γκούνερ Χόκμαρκ, που είναι ο εισηγητής μας για την οδηγία, για την ανάκαμψη και εξηγήση των τραπεζών. Ο κύριος Τόρβαλτς μίλησε για την πιθανότητα διαφορετικής μεταχείρισης των τραπεζών ανάλογα από το κράτος στο οποίο δραστηριοποιούνται και τη χρηματοπιστωτική του κατάσταση. δεν απαντήσατε συγκεκριμένα. Αλλά πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Γκούναρ Χόκμαρκ. Σας ευχαριστώ. Μας τελειώνει ο χρόνος. Είναι πολύ σημαντικό να σου πω, Μισελ, ότι ήσουν ανέκαθεν πρόθυμος για συζήτηση και έτοιμος να συμβάλεις ε, για να σημειωθεί πρόοδος και σε εκτιμούμε ιδιαίτερος γι' αυτό, γιατί πραγματικά βοήθησες με το επικοδομητικό σου και το ρεαλιστικό σου πνεύμα στην προώθηση της οδηγίας αυτής για την ανάκαμψη και την εξήγηση των τραπεζών που θα είναι ο κρογωνιαίος λίθος της Τραπεζικής Ένωσης ε, και σημαντική δική σου παρακαταθήκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η κατεξουδότηση πράξης να είναι σαφής και ασφαλής και να παραμένουν στο πλαίσιο για το οποίο έχουν αποφασιστεί. Γιατί μερικές ε, ομάδες προσπαθούν να επαναφέρουν κάτι που είχαμε χάσει στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό όμως να μείνουμε στην μέθοδο που συναποφασίσαμε με το Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση που θα πρέπει να στηρίζεται στην λήψη υπόψη και του μεγέθους των τραπεζών και την έννοια του κινδύνου. Θα πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος και με τον κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτή τη φόρμουλα θα πρέπει να την κρατήσουμε, γιατί την έχουμε συναποφασίσει. Και για να προχωρήσει η κατεξουσιοδότηση πράξη και να εγκριθεί εμπρόθεσμα, εγκαίρος, είναι σημαντικό να κρατήσουμε ε, απαράλλακτη την πορεία μας και να δείξουμε πυγμή στις διαπραγματεύσεις. Επίση για την παρακαταθήκη που μας αφήνεις, μας παρουσίασε πολλές νομοθετικές προτάσεις και μερικές φορές είχαμε και διαφορετικές απόψεις. Ε, πρόκειται για ένα τομέα που χαρακτηρίζεται από τον κίνδυνο και είναι δύσκολο να ληφθεί υπόψη πάντα, να συμπίπτουν οι απόψεις για τον κίνδυνο. Και μερικές φορές είχαμε αποκλίνωσες εκτιμήσεις, αλλά τελικά Έχουμε σημαντικά ε, νομοθετήματα, ΜΥΦΙΤ 2, τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει, ε, συστήματα ε, εγγύης καταθέσεων και την οδηγία για την ανάκαψη και την εξυγίαση. Αν θεωρήσουμε, όπως το πιστεύουμε, ότι έχεις, έχεις προχωρήσει πολύ στην νομοθεσία αυτή, θεωρήσω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η κατάσταση σήμερα, αν δεν ήσουν εδώ. Πιστεύεις ότι θα ήταν διαφορετική αν δεν είχαμε όλη αυτή την επιρροή από πλευρά σου. Ο κύριος ε, Πίτερ Σάιμον. Κύριε Επιτροπέ. Συγχαρητήρια και από πλευρά μου. Αυτή η τελευταία πενταετία είναι χαρακτηρισμένη από ζητήματα μακροχρόνια της διασφάλισης των καταθέσεων και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα και ήσασταν πάντοτε επικοδομητικός εταίρος, πάντοτε είχατε λύσεις να προτείνετε. Θέλω λοιπόν και προς τους συνεργάτες σας και, όλους, ε, και προς όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την επικοδομητική ατμόσφαιρα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη συμμετοχή, για την συμβολή τους σε αυτό το κοινό ε, Ταμείο Εκαθάριση, τον Γενικό Σα που είναι εδώ και που αύριο θα κάνουμε μαζί συζήτηση για τι λεπτομέρειε. Θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο θέλω να συζητήσουμε μαζί εσεί και εγώ. Γιατί μου φαίνεται ιδιαίτερα προβληματικό. Είπατε πολύ σωστά ότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τι ε, διεκδικήσει των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη, προκύπτει ότι οι τράπεζε ε, των οποίων η συνεισφορά ε, αντιστοιχεί στο 88% ή φτάνει μέχρι το 90% μπορεί να ε, καταβάλουν το 90% των συνεισφορών. Αυτό, εάν το αντιπαραβάλλουμε με το ερώτημα ε, του πώς αντιμετωπίζουμε τους μεγαλύτερους και πόσο αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο, εάν έχουμε αυτή την απόκληση μόνο 2% για τις μεγαλύτερες ε, τράπεζες, που θα καταβάλουν εάν αυξηθεί ο παράγων κινδύνου. Αυτό είναι νομίζω μικρό ποσοστό, αν το δούμε αυτόνομα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική διάσταση εάν υλοποιούνταν αυτό που τις τελευταίες ημέρες συζητείτε, εάν δηλαδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα με παράγωγα, γιατί η κατάσταση είναι ότι έχουμε μεγάλη επιβάρυνση για τις μεγάλες τράπεζες, εκεί που έχουμε μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο, έχουμε μια λύση για τις πολύ μικρές τράπεζες ή τις μικρές, τι γίνεται όμως εάν επιτρέψουμε να υπολογιστούν και τα παραγωγά με επιβάρυνση κατά 30% των ισολογισμών των μεγάλων τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν οι μεγάλες τράπεζες θα μπορούσαν απλούστερα απλούστατα να υποβαθμίσουν την ε, συμβολή τους. Και άρα πολλές μεγάλες τράπεζες, αν αναγνώσκω σωστά την κατάσταση, θα έμπαιναν στον, στην κατηγορία των μεσαίων ιδρυμάτων. Αυτό λοιπόν νομίζω έχουμε τον κίνδυνο να δούμε να υλοποιείται και να ανατρέπει όλο το σχεδιασμό μας το σχετικό με τον κίνδυνο. Θα ήθελα τη δική σας λοιπόν εκτίμηση γιατί είναι μια συζήτηση που τις τελευταίες μέρες φαίνεται να, να διαρρέει και από το Συμβούλιο. Ο κύριος Βάλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο θερμά για την εξαιρετική συνεργασία τα τελευταία χρόνια που θεωρώ ότι μπορούμε να σας χαρακτηρίσουμε ως προς τη συνεργασία σας με το Κοινοβούλιο ως ένα πραγματικό gentleman όλα αυτά τα χρόνια για όλα τα θέματα, το Insolvency 2, το την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξηγήση τραπεζών. Όλα αυτά λοιπόν. Είπατε ότι πρόκειται να υποβληθούν νέε προτάσει. Νομίζω όμω ότι πια είναι η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει τι προτάσει γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρειαστεί και τους έξι μήνες κατά πάσα πιθανότητα. Η πάση περιπτώσει μπορεί να διεκδικήσει τους έξι μήνες. Άρα πάμε για το Μάρτιο, 31 Μαρτίου του 2015 από σήμερα και μια και ο Οκτώβριο έχει 31 ημέρες. Θα ήθελα να παρακαλέσω στις αρχές του μηνός μάλλον και όχι προς τα τέλη να δούμε τις προτάσεις αυτές. Πολύ σημαντικό βεβαίως είναι να έχουμε ώστε όσο το δυνατόν πιο αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, να μην τεθεί το χρονοδιάγραμμα και επίσης Θέλουμε και τη διατήρηση των εγγύσεων και τη σταθερότητα, και κυρίως για τα μακροπρόθεσμα ε, μέσα αλλά και τη διαχείριση του κινδύνου και την υποχρέωση ενημέρωσης. Τα νομοθετήματα νομίζω θα είναι συμπλήρωση όλων αυτών που ισχύουν τώρα και εν τέλει θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε, να, να... θα πρέπει πολύ προσεκτικά να το δηλώσουμε αυτό και να το καταφέρουμε, θα πρέπει να παραμένουν συνεπείως προς την οδηγία. Η διάρθρωση του κινδύνου όχι μόνο για τον τομέα της ασφάλειας αλλά και για τη CDF4 για τον τομέα των τραπεζών θα πρέπει να εξεταστεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Επίτροπε και εσείς αλλά και η εποπτική αρχή να ακολουθήσει μια πολύ αυστηρή επιλογή και δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέρνερ Λάγκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου στις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια. Μαζί περάσαμε πέντε χρόνια μαζί με τον πρώην συνάδελφο Μισελ Μπαρνιέ σε μια εξαιρετική συνεργασία που μπορεί να αποτελέσει νομίζω πρότυπο για άλλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Από την άλλη διαπιστώνουμε ότι το όλο εγχείρημα της ε, ρύθμισης του τραπεζικού τομέα αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τους διάφορους παράγοντες και κυρίως ε, τα κράτη-μέλη όπου βλέπουμε ότι ορισμένες λεπτομέρειες δεν θέλουν να τις δεχθούν όπως είχαν υποσχεθεί όσον αφορά τη διεθνή διάσταση τώρα. Πριν από τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε με, τη, με την ε, ρύθμιση των παραγόγων με 19 πράξεις κατά εξουδοδότηση, ε, εκ των οποίων την πρώτη, η πρώτη ήταν πολύ διαφιλονικούμενη, αλλά πέρασε. Μετά είχαμε τις ενδιάμεσες εκλογές, το midterm στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν έφεραν τα αναμενόμενα για μας τουλάχιστον αποτελέσματα και τώρα έχουμε πάλι mid-term elections. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αυτές οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τη ρύθμιση των παραγόγων μπορούν να προχωρήσουν ή όχι και επίσης για μια λεπτομέρεια ουσίας όμως, γιατί είχαμε αποφασίσει τα παράγωγα που έχουν σταθεί στο ε, χρηματιστήριο να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερο τρόπο, αλλά δεν έχουν αποκλειστεί ακόμα από τα χρηματιστήρια των Ευρωπαϊκών κρατών. Είχαμε συμφωνήσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κατέθεται ένα κατάλογο των ε, χρηματιστηρίων τρίτων κρατών, αντίστοιχο με αυτό ε, των ΗΠΑ, δηλαδή που εξαιρούνται από την αμοιβαία υποχρέωση συναλλαγματική ισοτιμία, εκεί δηλαδή που η πραγματική οικονομία μπορεί να επηρεαστεί από αυτά τα ε, παραγωγά. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν κύριε Επίτροπε, αν, βλέπετε, αν διαβλέπετε κάποια δυνατότητα, αυτός ο κατάλογος που μας, είχε υποσχεθεί, μας είχατε υποσχεθεί και στη τελευταία ανάλυση είναι κομμάτι της νομοθεσίας. Εάν πιστεύετε λοιπόν, αν μπορείτε να μας δώσετε δέσμευση, ότι πρόκειται να δημοσιευθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ε, εκτίμηση και το θαυμασμό μου για το τιτάνιο έργο των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπό την καθοδήγηση του Επιτρόπου Μισελ Μπαρνιέ. Και έχω δύο σύντομες ερωτήσεις ή σχόλια για τον κανονισμό με τα μέτρα επίπεδου 2 σε ό,τι αφορά τον νέο μηχανισμό εξυγίασης και την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίαση των ε, τραπεζών. Ε, το θέμα των εισφορών στο Ταμείο είναι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα σημαντικά. Το θέμα είναι ε, η συμμετοχή στο σύστημα ε, θεσμικής προστασίας. Είναι σημαντικός ε, παράγον μείωσης ή μετριασμού του κινδύνου και θα είναι σημαντικό, σημαντική επιρροή της στην εκτίμηση κινδύνων για γραία και μεσαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, ε, η, ομάδα για τις ε, υποχρεώσεις ε, για το αποθετικό και η μείωση τη, της ομάδας αυτής, η μείωση του αριθμού των μελών και θα είπατε θα εφαρμόζεται μόνο σε τραπεζικούς ομίλους και όχι σε κάποιες συνεταιριστικέ τράπεζε, ε, που είναι μικρότερα, μικροπιστωτικά ιδρύματα, αλλά συμμετέχουν σε ένα δίκτυο. Μήπω θα μπορούσαν και αυτά, ε, τα, αυτές οι μικρότερες τράπεζες που συμμετέχουν σε δίκτυο να τη χάνουν εξαίρεση για να μην βρεθούν σε, σε δυσμενή θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσει. Και τελευταίος ο μιλητής, παρακαλώ, σύντομη ερώτηση από τον κύριο Σβέν Γκίγκολτ. Ε, αγαπητή Μισελ Μπαρνιέ. Ευχαριστώ και εγώ για την ανέκαθεν καρποφόρα και θερμή συνεργασία. Και Ελπίζα να μείνετε λίγο περισσότερε θέσει, γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Χίλ θα σα διαδεχτεί επάξια. Ίσως Χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο ο πρόεδρος Γιούνκερ για να ξανασκεφτεί τις προτάσεις του και να τις ε, προσαρμόσει ενδεχομένω. Έχω πέρα του, του, του σχολείου και μία ερώτηση. Στο σχέδιο ε, κατεξοδότηση πράξης για τη θεραγκαιότητα 2 που κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό στα διάφορα λόμπι βλέπουμε ότι τα προγράμματα ε, η κατανομή των προγραμμάτων ε, από τίτλου που προέρχονται από τυλοποίηση έχει αλλάξει. Πέρασε από το τριπλό Β, ε, ABC με τριπλό Β, σε ένα πολλαπλασιαστού και 17% και μετά με επεμβάσεις των κρατών μελών ξαφνικά η κατανομή του κινδύνου έπεσε στο 8,5% και τελικά η Γενική Διεύθυνση Εκφήν ζήτησε περαιτέρω μείωση και καταλήξαμε στο 5% σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή μειώθηκε κατά πολύ ο παράγων κίνδυνος. Και η ΑΙΟΠΑ είχε δώσει τελείως διαφορετικά στοιχεία στην αρχή. Πού στηριχθήκατε για να μειώσετε τον πολλαπλασιαστή κινδύνο και να το μειώσετε τόσο σημαντικά τι στοιχεία στηριχθήκατε. Αν δεν είστε έτοιμο να απαντήσετε τώρα, θα ήθελα να μου στείλετε γραπτή εντύπωση ποια είναι η εμπειρική βάση για την ε, ευνίδια μείωση του πολλαπλασιαστού κινδύνου για τα προϊόντα τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση, τον ε, ABS δηλαδή. Ευχαριστώ, ο κύριος Παρνιά. Για το θέμα που παρέλειψε προηγουμένως, την ερώτηση δηλαδή για το κατά πόσο μπορεί να γίνει έκπτωση των φόρων ανάλογα με το κράτος μέλος. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε, αλλά ακόμη δεν το έχουμε λύσει. Να αποφευθεί η διπλή φορολόγηση, δηλαδή. Αυτή ήταν η μέρημνα του συναδέλφου. Πάντως, με τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΤ και με τη Γενική Διεύθυνση ΓΙΟΥΡΙ ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, αναζητώντας την καλύτερη λύση για να αποφύγουμε τη διπλή φορολογία. Γκίναρ Χακμαρκ. Θερμά ευχαριστώ για την αγαστή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα και φυσικά έχετε και την ε, έκθεση για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών. Σας διαβεβαιώ, όπως είναι και καθήκον μου άλλωστε, ότι θα παραμείνουμε πιστοί στα κείμενα του επίπεδου 1 και υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επίσης ε, επαγρυπνεί για τα θέματα αυτά. Και φυσικά οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τη θέληση των δύο πτυχών της νομοθετικής αρχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραγωνίσουμε, δεν θα αποφύγουμε ή δεν θα παραμορφώσουμε τα κείμενα του επίπεδου 1 με τις της πράξεις και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Βέβαια, έχουμε την υποχρέωση, με βάση την εντολή μας και το έργο που μας έχει ανατεθεί, έχουμε την υποχρέωση στις καταξιδότητες πράξεις ε, να καταστήσουμε εφαρμόσιμα και λειτουργικά τα κείμενα συγκεκριμενοποιώντα μερικά θέματα και λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε του τραπεζικού τομέα και των τομέα των ε, ασφαλιών. Τώρα, ποιος είναι ο κίνδυνος με βάση την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα και την πορεία μας. Φυσικά στόχος δεν είναι η πλήρης απάλληψη των κινδύνων. Είναι αδύνατο στον τομέα αυτό, σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, να απαλείψουμε πλήρως τον, κίνδυνο. Απλώς θέλουμε να γνωρίσουμε τον κίνδυνο ώστε να προλάβουμε κάποιους κινδύνους, να τους ελέγξουμε και να προβλέψουμε κάποιες εγγυήσεις όπου είναι απαραίτητο. Και στην οικολογία αλλά και στην οικονομία η πρόληψη ε, στοιχίζει πολύ λιγότερο από τη θεραπεία ή την επιδιόρθωση. Και ακόμη και σε περίπτωση θεραπείας και επιδιόρθωσης θα πρέπει και εκεί να είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί καλύτερα είναι ελεγχόμενοι η αναμενόμενη θεραπεία παρά να είναι άτακτη ή αυτοσχέδια και να γίνεται σπασμωδικά την τελευταία στιγμή όπως έγινε μερικές φορές με την κρίση. Θέλουμε τα κείμενα να εφαρμοστούν, οι κατεξουσίδωτοι πράξεις να εγκριθούν και να καταστήσουν λειτουργικά τα κείμενα. Είναι περίπλοκος ο κλάδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η εποπτική λειτουργία. Φυσικά τώρα που τα κείμενα έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί και είναι γνωστά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη ρήτρα αναθεώρησης Γκέρνερ, που έχουμε προβλέψει σε πολλά από τα κείμενα αυτά. Και στη νέα φάση ρύθμιση που θα περάσουμε δεν θα ε, ξανακάνουμε τα ίδια, δεν θα επαναλάβουμε το ίδιο έργο. Θα δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες, πού υπάρχουν κενά, πού θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συμπεριφορές και στις νέες καταστάσεις και όπως είπα και προηγουμένως ε, θα πρέπει με τον πιο αντικειμενικό τρόπο να αναζητήσουμε τα, τις αδυναμίες και να τις συμπληρώσουμε. Τα κείμενα είναι απαραίτητα πραγματικά, είναι πολύ σημαντικά και η ιδέα το να έχει η Ευρώπη μέσα μέσω μιας, νέας, μέσω μιας καινούριας ή υπάρχουσας αρχής την ικανότητα να επιβάλλει κυρώσεις, πρόστιμα σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διακυβεύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι κάτι καινούριο. Και θα μας προβληματίσει και στο μέλλον. Ο Σάιμον μίλησε για το θέμα της αναλογικότητας, τη λήψη υπόψη του μεγέθους, του ρόλου και του βάρους των επιχειρήσεων. Αυτό το κάναμε. Και από τα στοιχεία που σας έδωσα είδατε ότι οι μεγάλες τράπεζες οι τράπεζες που έχουν και το μεγαλύτερο τμήμα του ενεργητικού θα καταβάλουν και τις μεγαλύτερες φορές και θα περικοδοτήσουν το Ταμείο Εξυγίασης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιπλοκότητα της έκθεσης των παραγωγών, οι μεγάλες τράπεζες θα, θα καταβάλουν πάνω από το 90% των εισφορών, οι μέσες τράπεζες 9% και οι πιο μικρές τράπεζες 1% του προϋπολογισμού του Ταμείου Εξυγίασης. Με αυτά τα ποσοστά και στοιχεία εργαζόμαστε. Τώρα, ο Πίτερ έθεσε μια ερώτηση για τα παράγωγα. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν για τις τράπεζες, τις μικρές τράπεζες. Ε, δεν έχουμε εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες. Αυτό οδηγεί σε ε, με, σε διακύμαση των παραγόγων ε, μεταξύ των τραπεζών ή μεταξύ των διαφόρων χωρών για το ίδιο ποσοστό. Και για να εξασφαλίσουμε σε μια εναρμόνιση των παραγόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να έχουμε μια μακροπροληπτική μεταχείριση του της μόχλευσης του κινδύνου, όπως προβλέπεται στην ε, τέταρτη δική και τις κεφαλαϊκές ε, απαιτήσει και να εφαρμόζεται και στα παράγωγα τουλάχιστον όταν εξετάζουμε τις αιτήσιες εισφορές. Και, και αύριο φαντάζομαι θα συνεχίσετε με το Γενικό Διευθυντή τη συζήτηση. Θα μπορούσαμε να βρούμε συμβαστική λύση μεταξύ μιας αμυγίους εφαρμογής του λογιστικού, των λογιστικών κανόνων και της εφαρμογής της προληπτικής εποπτείας, όπως προβλέπει η Οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Μία ερώτηση αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και για τη φερεγκιότητα 2 και για την τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Ε, για να σας παρουσιάσουμε αυτά τα κείμενα το συντομότερο δυνατόν, παρόλο που είναι περίπλοκα και πολυσύνθετα. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε και το χρόνο της διαβούλευσης και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα Ελπίζουμε ήδη από τον Οκτώβριο να σας υποβάλουμε αυτά τα δύο κείμενα και ελπίζω να έχουμε και συνεργασία με το Συμβούλιο για να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Πάντως, για νομικούς λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να ελέγξω, δεν αποκλείεται η κατεξοδότηση πράξη να υποβληθεί επίσημα τον Νοέμβριο. Πάντως, φροντίζουμε να είναι συνεκτικά τα κείμενα μεταξύ τους. Ευχαριστώ και τον Βέρνερ Λάγκεν για τη συνεργασία μας και το πολύ σημαντικό έργο. Τον ευχαριστώ για τη φιλία του και την εμπιστοσύνη του που μας στήριξαν πολύ. Σε ό,τι αφορά τα παράγωγα, ε, για συζητήσεις που έχουμε τους Αμερικανούς για την ισοδυναμία, με εμπιστοσύνη αλλά χωρίς αφέλεια, είπα και προηγουμένως. Πρόσφατα μίλησα με τον Tim Assad, τον νέο αρμόδιο για την CFTC. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τηλεφωνική συνομιλία και είχαμε ε, και απεσταλμένους μας στην Ουάσιγκτον για προσωπικές συνομιλίες και ο κατάλογος αυτός ε, θα δημοσιευθεί, τον επεξεργαζόμαστε και η μεν και η δε. Θέλουμε, θα θέλαμε ένα, μια συμφωνία με τους Αμερικανούς και με τη CFTC και πριν το τέλος της δικής μου θητείας, ή δυνατόν. Δανούτα Χιούμπνερ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αναφέρθηκατε στο θέμα της, του αποκλεισμού της εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις ε, των μελών του ίδιου IPS ή του, των μελών του ίδιου συστήματος αμοιβαίων εγγύσεων. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αρκεί η λειτουργία του IPS να οδηγεί σε διασύνδεση των μελών του IPS παρόμοια με αυτή ενός τραπεζικού ομίλου. Θα συνεχίσετε αύριο τη συζήτηση με τον Ολιβία για το θέμα αυτό. Θέλουμε μια συγκεκριμένη και σαφή διατύπωση για το θέμα αυτό. Επίσης για την, για την εξαίρεση των εκθέσεων μεταξύ των ομίλων θα είναι της τάξης του 10% και κατά τη γνώμη μας αυτή, αυτός ο αποκλεισμός, αυτή η εξαίρεση 10% θα ευνοήσει κατά τη γνώμη περισσότερο τις μεγάλες και όχι τις μικρές τράπεζες. Πάντως είπα ότι όλες οι αποφάσεις μας στόχο είχαν να διευκολύνουν τις μικρές τράπεζες και τα μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι να τα επιβαρύνουν γραφειοκρατικά και κυρίως τις, τους συνεταιρισμούς, συνεταιριστικές τράπεζες που ανέφερες και εσύ Ντανούτα. Σβέν Γκίγκολτ, σε ευχαριστώ και σένα και για την αξιολόγηση και τα καλά σου λόγια. Δεν θα ξεκινήσουμε συζήτηση για τη μελλοντική σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ενθαρρύνουμε στα πλαίσια του, της Φερικιώτας 2 μια τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας. Και αυτό Φαίνεται και από την παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σας τα εξήγησε και ο κύριος Δράγκη πριν από λίγο για να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Με τα νέα μέλη της Επιτροπής θα εξετάσετε ένα επενδυτικό σχέδιο και εκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διαδραματίσει το ρόλο της γιατί πιστεύω ότι με την ομοθεσία μας θα πρέπει συνειδητά και σοβαρά με τις απαραίτητες προφυλάξεις βέβαια να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε ε, την χρηματοδότηση της οικονομίας και η υψηλής ποιότητας τυλοποίηση, όπως αυτή που επεξεργαζόμαστε και θα προτείνουμε, θα πρέπει να συμβάλλει ε, σε, με μια διαφανή και υγιή τυλοποίηση υψηλών προδιαγραφών, θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Φυσικά χρησιμοποιούμε ως βάση το έργο της ΑΙΟΠΑ και τις άλλες δύο εποπτικές αρχές. Έτσι κάνουμε ε, μια τεχνική κατανομή, ένα πολύ εκλεπτισμένο έργο κατανομής και βαθμονόμησης. Και μάλιστα ο Μπεράρ εδώ ήταν στο πλευρό μου και στο Συμβούλιο Υπουργών του Μιλάνου. Και άκουσε και τους υπουργούς. Γιατί και οι υπουργοί ξέρουν για την οικονομία της χώρας τους και είναι και αυτή υπέρ της τιτλοποίησης υψηλής ποιότητας. Και μεταξύ αυτών των δύο ορίων θα κινηθούμε. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπαρνιέ. Really, Σας ευχαριστούμε και για την παρουσία σας και για το έργο σας κατά τη διάρκεια της θητείας σας και ελπίζω να μην χάσουμε την επαφή μας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την κατεξοδότηση πράξης αύριο στις 5. Έχουμε και μία νέα ιστοσελίδα που δίνει πρόσβαση σε όλες τις κατεξοδότησεις, κατεξοδότηση πράξης και τα εκτελεστικά ε, ε, μέτρα καθώς και τα συναφή έγγραφα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Λύεται η συνεδρίαση.